So, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Yeah. ο πρόεδρος θα έρθει λίγο αργότερα, γι' αυτό και αναλαμβάνω εγώ να κήρυξω την έναρξη της συνεδριάσεως σήμερα. Καλημέρα σας και παρακαλώ, ε, κλείστε το στόμα σας. Κλείστε το. Δύο. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θα έχουμε έναν, ε, μια κάμερα της ΙΤΕΚ σήμερα εδώ που θα κάνει γυρίσματα για ένα μεγαλύτερο ε, πρόγραμμα καταγραφής των εργασιών του Κοινοβουλίου. Θα παίρνει λοιπόν εικόνα αλλά όχι ήχο, να ξέρετε. Σημείο 3. Έχω εγώ την ε, έκθεση η οποία αφορά την εξέλιξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Πού είμαι, πού το έχω. Όχι αυτό. Είναι για το 4. Λοιπόν, στο 3 μπορώ να σας ενημερώσω ότι ο τριμερής διάλογος CRDCR ε, που έχω αναλάβει ο συγητής έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες μέτρα για την καταπολέμηση της νομοποίησης των μεγάλων εκθέσεων και ούτω καθεξής αντιμετωπίστηκαν. Προσεχής τριμερής 7 Νοεμβρίου. Για το ΕΜΙΡ και την αναδιατύπωση της οδηγίας ΕΜΙΡ. 12 Οκτωβρίου συμφώνησαν οι συνομοθέτες την άρση της υποχρέωσης εκαθάρισης αλλά θα γίνει συζήτηση για την καθάριση στα ασφαλιστικά ταμεία και για, τους, για τον περιορισμό των κινδύνων. Η υποχρέωση λογοδοσία στο πλαίσιο του, της νομοθεσίας αυτής είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε γιατί δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε χρόνος. Ε, έχουν μείνει σε τεχνικό επίπεδο αρκετά ζητήματα να διατυπωθούν από τεχνική ομάδα. Πανευρωπαϊκό προϊόν, εξωτερικό προϊόν πανευρωπαϊκό. 11 Οκτωβρίου πρώτος τριμερής θεσμική ανταλλαγή απόψεων πεδίο πιθανών συμβασμών σε σχέση με την αδειοδότηση, τους παρόχους το, που μπορούν να προσφέρουν το προϊόν, τους εφαρμοστέους κανόνες, την ε, εναλλαγή και η τεχνική συνεδρίες, τεχνικές συνεδρίες να λαμβάνουν, να ετοιμάσουν κείμενα για τον προσεχή στις 25. Τελευταίο. Έδρα έμπα. Ότ Μαρκάρας, Πέγμος Περές, εισηγητές. Στις 17 Οκτωβρίου επιβεβαίωσε το Κορεπέρ την πολιτική συμφωνία για την έδρα της ΕΜΠΑ και κυρίως τα λοιπά πολιτικά ζητήματα και με βάση μια κοινή δήλωση και προσέγγιση για την τοποθέτηση έδρων των υποκεντρωμένων υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2019. Ξαναγίνεται η διαβούλευση με την ΕΚΟΝ στο πλαίσιο λοιπόν διοργανικών διαπραγματεύσεων. Και να ακόμα ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει. Τριμερής διάλογος BRRT είναι τα υπόλοιπα του CRD-CRR. Κομμάτι της ε, διαβούλευση για τα τραπεζικά. Εχθές έγινε η συζήτηση στον τριμερή διάλογο με αρκετή πρόοδο για την επίλυση ζητημάτων όπως δομημένων ομολόγων, ε, ε, συνεταιριστικών δομών κτλ. Ε, υπαγωγή στην ε, δικαιοδοσία τρίτων χωρών και άλλα ζητήματα. Πρόοδος επιτεύχθη ως προς την αναγνώριση των διαφορών στις θέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Προσεχής τριμερής στις 6 Νοεμβρίου. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει ο διάλογο, ο ε, διάλογο για την BRRD και υπό την έννοια της ε, CDR, διότι έχουν μπει ε, σε ένα είδο ομοιρίας στα δύο αυτά ζητήματα τη οδηγία και του κανονισμού σε σχέση με την BRRD. Όσο δεν προχωρά δηλαδή η BRRD δεν μπορούμε να έχουμε ουσιώδη πρόοδο στα θέματα CRD-CRR, γιατί το Συμβούλιο παρεμποδίζει η αδίποτε πρόοδο. Ευχαριστώ λοιπόν και προχωρώ στο σημείο 4. με τη δική μου έκθεση. Εφαρμογή νομικών διατάξεων και κοινή δήλωση για την κοινοβουλευτική εποπτεία αποκεντρωμένων ε, ε, υπηρεσιών και συνεχίζω στα γερμανικά. Στη γνωμοδότηση αυτή λοιπόν προς την ΕΚΟ, ΕΚΟΝ μια κοινή γνωμοδότηση για τις αποκεντρωμένες οδηγίες προς, ε, υπηρεσίες προς την ΑΦΚΟ με αρμόδιο γνωμοδότηση στον κύριο Σόπφλιν ε, και προχωρώ στην αναφορά ότι στις 26 Σεπτεμβρίου απεστάλλει η γνωμοδότησή μου 1500 μόνο στοιχεία έχω δικαίωμα να διατυπώσω, επομένως είναι πολύ σύντομη η γνωμοδότηση προς την ΑΦΚΟ 25 Οκτωβρίου λίγη ακριβώς 7 μέρες δηλαδή ε, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών ε, και 19 ή 20 Νοεμβρίου θα γίνει η συζήτησή τους στις 21 ή 22 Ιανουαρίου πλέον εδώ στην Επιτροπή των Οικονομικών θα γίνει ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες ε, που έχουν στενή, στενή συνάφεια με την ε, Επιτροπή μας είναι η ΕΣΜΑ, η ΕΜΠΑ, η ΑΙΟΠΑ, η SRB. Τα λοιπά θα τα δείτε στη γνωμοδότησή μου. Την έχετε λάβει. Καταρχάς γίνεται μια μνήμα στις ε, υποχρεώσει στα καθήκοντα των αποκεντρωμένων οργανισμών, ότι πρέπει να ασκούν πλήρως και εμπροθέσμως όλα τα καθήκοντα που απορρέμουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο και να μην υπερβαίνουν τις εντολές που τους έχουν δοθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης, ε, λέμε ότι θα πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και να εφαρμόζουν τι αρχέ τη βελτίωση νομοθετικού έργου ε, πλήρω, ιδιαίτερω μέσω διεξαγωγή ανοιχτών δημόσιων διαβουλεύσεων όσον αφορά τα σχέδια προτάσεων για δευτερογενεί και τριτογενεί νομοθετικέ πράξει. Επίση αναφερόμαστε στην πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου σε συνεδριάσεις εποπτικών συμβουλίων και ομάδων ενδιαφερμένων σε επίπεδο οργανισμών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν αυτοί στα εποπτικά συμβούλια, που είναι τα κύρια ε, όργανα λήψη αποφάσεων, αλλά και σε συνεδριάσεις ε, με εκπροσώπους των οργανισμών που θα επέτρεπαν την διευκόλυνση του τρόπου λήψη αποφάσεων, της αντίληψης ε, για τον τρόπο λήψη αποφάσεων. Συμμετοχή λοιπόν στα όργανα αυτά για το Κοινοβούλιο θα σήμαινε καλύτερη κατανόηση και επιτάχυνση των εργασιών. Το Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων συστηματικά και σε ισότιμη βάση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο κριτήρια σε σχέση με τον τόπο εγκατάσταση όλων των οργάνων λοιπόν και όλων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, διαμορφώνονται συστηματικά και σε ισότιμη βάση από το Κοινοβούλιο μαζί με, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι έχουμε κατώτερο καθεστώς, χρειάζεται να μας αναγνωστεί ισότιμη συμμετοχή με το Συμβουλίο και την Επιτροπή στο καθορισμό και τη σταθμίση των κριτήριων. Επίσης τονίζω με την γνωμοδότηση ότι ο τόπος εγκατάστασης ενδέχεται να καταστεί δυνατή μια κοινή διοικητική στήριξη, κοινέ υπηρεσίε διαχείριση εγκαταστάσεων μεταξύ των οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει αυτό να επηρεαστεί. Ε, το τονίζουμε λοιπόν ε, και στην ε, γνωμοδότηση ότι η άσκηση εξουσιών και καθηκόντων, δομή διακυβέρνηση κτλ. βασική χρηματοδότηση δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον τόπο στον οποίο αυτό ο οργανισμό είναι εγκατεστημένο και πρέπει αντιθέτω ή δυνατόν, όπου είναι δυνατόν, να προβλεφθεί μια κοινή διοικητική στήριξη και κοινέ υπηρεσίε διαχείριση. Αυτά για τη γνωμοδότησή μου. Προ το Κοινοβούλιο. Ο Brian Hayes είναι ο σκιώδης ηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ. Δεν τον βλέπω εδώ, ούτε βλέπω να τον εκπροσωπεί κανείς. ECR. Η κυρία Σουίνμπερν σκιώδης, αλλά ούτε αυτή είναι εδώ, ούτε και βλέπω να αντικαθιστά κανείς από το ECR. Λίμπε. Α, ε, συγγνώμη, η κυρία Βίρινγκ εκ μέρους της Άλντε είναι εδώ. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κύριε Σίμωνα για το σχέδιο αγνομοδότησης που είναι συνοπτικό εύστοχο και επικεντρώνεται στα ουσιώδη. Ε, δηλαδή, στόχος μας είναι να δώσουμε μια σαφή εικόνα για το πώς θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών και των θεσμικών οργάνων μας, κυρίως α, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να δράσουμε στα πλαίσια και στα όρια της εντολής που έχουν οι οργανισμοί και θα πρέπει να τα ξεπερνούν. Συμφωνώ πάντως με τον εισηγητή ότι είναι σημαντικό να οργανώσουμε την δυνατότητα και σε άλλους ενδιαφερόμενους να δίνουν τη γνώμη τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να αυξηθεί η επικοινωνία πριν, κατά και μετά τη δημιουργία δευτερογενούς και τριτογενούς νομοθεσίας. Συμφωνώ με το μήνυμα του Συμβουλίου ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ισότιμο βάρος με το Συμβούλιο, Συμβούλιο κατά την απόφαση του τόπου έδρας ε, της κύριας έδρας ε, του κάθε οργανισμού. Συμφωνώ λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε ε, συνομοθέτες ε, και ο οίκος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, έξω και το αίτημά μας που είναι πολύ θεμητό κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Γουαλτιέρη. Δεν βλέπω εκπροσώπους ούτε των πρασίνων. Περβάς, ήθελε το λόγο. Ούτε από την ΚΟΕ κανένας, οπότε περνάμε στο Catch the Eye, Ευχαριστούμε τον εισηγητή που κήρυξε το εναρκτήριο λάκτισμα της συζήτησης. Άλλωστε, η συζήτηση ουσιαστικά ξεκίνησε από προηγούμενη έκθεση. Και ο λόγος που η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει επιληφθεί του θέματος είναι ακριβώς γιατί ε, ζήσαμε το επώδυνο θέμα της ε, μετεγκατάστασης του οργανισμού φαρμάκων ή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, που και αυτή έπρεπε να αλλάξει έδρα. Εξού και η, το αίτημα αναθεώρησης, που συμπίπτει με μία από τις ένα από τα συμπεράσματα της συμφωνίας μας με το Συμβούλιο. Οπότε, ε, ξεκινάμε τη συζήτηση με βάση ε, κάτι που γνωρίζουμε και είναι και αρμοδιότητά μας, το θέμα της λειτουργίας των οργανισμών και θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε και κάποια διδάγματα από τις γνώσεις μας μέχρι τώρα. Καταρχήν στην κοινή δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι η έδρα των οργανισμών θα εμπίπτει στη συναπόφαση και θα περιλαμβάνεται στη βασική νομοθεσία, όπως γίνεται για τους οργανισμούς μας και που δεν ισχύει για τα άλλα θέματα. Και σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να επιμείνουμε ότι ο καθορισμό ε, των εδρών των οργανισμών εμπίπτει στη συναπόφαση. Σε ό,τι αφορά τα μέσα των οργανισμών. Αν έχουμε διοργανική δήλωση για το θέμα αυτό, θα πρέπει στη δήλωση να δεσμεύονται τα θεσμικά όργανα να εφοδιάζουν ε, με τον κατάλληλο προπολογισμό του οργανισμού για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο του. Επίση, θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή μα να εξετάσει το περιεχόμενο τη δήλωση για τη διακυβέρνηση των οργανισμών. Γιατί βλέπουμε ότι στη δήλωση Υπάρχουν κάποια αναλυτικά σχόλια για τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, για τη σύνθεση των εκτελεστικών συμβουλίων και να ε, θυμίζω ότι για τα εκτελεστικά στελέχη αναφέρεται ότι ο διοικητής του οργανισμού κάνει τη στελέχωση του επιτελείου του, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου όχι μόνο ο ο διοικητή θα περάσει τη διαδικασία έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι που ισχύει για το, Ευρωπα... Ε, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίαση, το SRB. Οπότε πιστεύω ότι εμεί έχουμε εμπειρογνωμοσύνη και μπορούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση, να την τροφοδοτήσουμε και να διευρύνουμε τη δήλωση που είναι κάπως περιοριστική σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση των οργανισμών. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σίμων. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο τοποθετήσεις. Βεβαίως και περιμένω τις ε, τροπολογίες παιδόνς. Όπως είπα και πάλι, μέσα στις επόμενες 7 ημέρες, 25 Οκτωβρίου δηλαδή, λίγη η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Exactly. 25 Όντως, 25 Οκτωβρίου το μεσημέρι. 19 και 20 Νευρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ στις 21 και 22 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο θέμα, στα επόμενα θέματα για την ακρίβεια, το 5 και το 6 καλυμμένα ομόλογα και δημόσια υποπτία των καλυμμένων ομολόγων και ανοίγματα με τη μορφή των καλυμμένων ομολόγων. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Μπέρντ Λούκε, που έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κοιόδης συγγετές... για την πολύ καλή συνεργασία και τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει. Νομίζω ότι είμαστε στον ε, πολύ καλό δρόμο να ολοκληρώσουμε αυτές τις δύο προτάσεις εκ μέρους της Επιτροπής μας, εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Η εντύπωση που έχω αποκομίσει μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία στα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε πιο εντατικά και ίσως υπάρχουν ακόμη κάποιες αποκλήσεις απόψεων. Ε, το ένα αφορά τον ορισμό των ε, επιτρεπτών εξασφαλίσεων για τα καλυμμένα ομόλογα. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι θέλουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ εκείνων που προβλέπονται ήδη στον ε, ΣΕΡΕΡ και που δίνουν προνομιακή μεταχείριση ε, από την ομοθεσία για τα καλυμμένα ομόλογα, αλλά και ότι θέλουμε ένα χωριστό άρθρο που θα δίνει ποιοτικό θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις ε, εξασφαλίσεις, αυτές τις εγγύησεις. Εδώ, στη διαχείριση κινδύνου, έχουμε αποκλήσει απόψεων σε σχέση με το πόσα θα πρέπει το ευρωπαϊκό, σε ποιο βαθμό θα πρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο να παρεμβαίνει με λεπτομέρειες. Θέλουμε βεβαίως μια ρύθμιση, μια οδηγία προσδιορίζω με αρχές, με προσδιορισμό αρχών που θα πρέπει να επιδιωχθούν, αλλά από την άλλη ε, θα πρέπει ίσως να απαιτήσουμε και μια ποιοτική διαμόρφωση του σύνθεσης των καλυμμένων ομολόγων, της διασφάλισής τους, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αυτή να υπονομευθεί. Επίσης ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με τα παράγωγα στις ε, δομές ομαδοποίησης για το αν μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν ε, για την αποτροπή κινδύνου και τι είδους μέτρα κάλυψης πρέπει να προβλεφθούν. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ακόμη με τους υγιτές και να καταλήξουμε ή τουλάχιστον να καταλήξω εγώ σε ένα συμπέρασμα γιατί βλέπω ότι έχουν διαφορετικές θέσεις οι ομάδες. Επίσης, στον κανονισμό η δυνατότητα επέκτασης ε, της, ε, του ληξιπρόθεσμου, της προθεσμίας δηλαδή. Υπάρχει μια πρόταση πρωτοβουλίας για την παράταση της διάρκειας ζωής και θέλουμε αυτή να την υπαγάγουμε στον όρο της ε, φερεγγιότητας, δηλαδή να την απαλλάξουμε από εξωγενείς παράγοντες. Πιστεύω ότι και στην οδηγία πρέπει να καταλήξουμε στην ίδια επιλογή και τελικά αυτό είναι ζήτημα αξιολόγηση του κινδύνου. Γιατί εάν η εκκίνηση του κινδύνου γίνει ανεξάρτητη από τη φερεγγιότητα, τότε η διπλή αυτή δυνατότητα, η διπλή προσφυγή προσφυγής δεν καλύπτεται. Η διπλή προσφυγή, ο μηχανισμός διπλής προσφυγής δεν καλύπτεται. Όπως θα έπρεπε. Και Μέχρι τώρα αυτή είναι η κατάσταση, όπως μπορώ εγώ να διαπιστώσω για τι συζητήσει που έχουμε κάνει. Περιμένω τις τροπολογίες βεβαίως των συναδέλφων από τις πολιτικές ομάδες και τις περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ και εκπροσωπώντας τον κύριο Ρωσάτη θα μιλήσει ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ. Είμαι Πολωνός. Ich bin ein Polen. Καταρχήν, ζητά συγγνώμη ο κύριο Ρωσάτη για την απουσία του. Μου ζήτησε να διαβάσω εκ μέρου κάποια σχόλια. Εκ μέρου λοιπόν του Δαρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέρνγκλου και τον εισηγητή και του σκιώδη εισηγητέ για το έργο του σε αυτή τη σημαντική έκθεση. Ο κύριο Ρωσάτη εκτιμά ότι τα περισσότερα μέλη ευθυγραμμίζονται με την αρχή ε, ε, την προσέγγιση επί των αρχών και θέλουν μια διαφάνεια στην αγορά καλυμμένων ομολόγων. Είναι εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία με του συναδέλφου και θα ήθελα να δώσω έμφαση σε κάποια σημεία παρόλα αυτά. Είναι υπέρ τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού σήματο που θα καλύπτει το καθεστώ για τα καλυμμένα ομόλογα και θα γίνεται διαφοροποίηση των καλυμμένων ομολόγων ανωτέρα ποιότητας από τα πιο επισφαλή μέσα. Ε, διευκρινίζει κάποιους ορισμούς ε, για το καλυμμένο ομόλογα και θέλει να ε, αλλάξει τον ορισμό για τους ειδικευμένου ε, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Επίσης, ε, δεν χρειάζεται να υπάρχουν ανώτατα όρια, γιατί χρησιμοποιούνται μόνο για μετριασμό κινδύνου, για την αντιστάθμιση κινδύνου τα καλυμμένα ομόλογα και ήδη εξασφαλίζουν επιπλέον προστασία στον κάτοχό τους κατά τη γνώμη του κυρίου Ρωσάτη θα πρέπει να υπολογίζονται με μία βάση καθαρής ταμιακή ροή. Επίσης, ο κύριος Ρωσάτη χαίρεται για την παράταση κατά μία διετία της ε, περίοδου της μεταβατικής για να μπορέσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές να προσαρμοστούν στην, ένο, στην Παρ' όλα αυτά, ε, θεωρεί ότι είναι πολύ επικοδομητική συνεργασία και στη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών παρ' όλα αυτά αναδείχθηκαν πολλές εκκρεμότητες, όπως το άρθρο 6α, 8 και 10 που χρήζουν περαιτέρω συζήτηση. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, ελαστικότητας και της τυποποίησης που χρειάζεται επίσης. Θέλουμε υψηλά πρότυπα για την αγορά καλυμμένων ομολόγων και ταυτόχρονα δεν θέλουμε να, διαφ... να ε, θέσουμε ένα αφιβόλιο να διακινδυνεύσουμε κάποια ευρύθυμα συστήματα και αγορές καλυμμένων ομολόγων. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ανάλογα και δικαιολογημένα. Ε, ε, θέλουμε τα soft bullets ε, για τους συντελεστές στάθμης κινδύνου και παράταση της λεκτότητας για να έχουμε μια εναλλακτική λύση και να επιτρέψουμε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο και να αυξήσουν την προστασία του επενδυτή. Βέβαια, οι λεπτομεριακές διατάξεις για την παράταση της λεκτότητας θα πρέπει να ρυθμιστούν και να προστατευτούν τα επενδυτικά συμφέροντα. Δεν είμαι υπέρ Αλλαγή τη κεφαλ... της δομής για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί δεν έχει γίνει αναλυτική ε, εξέταση. Πάντως, ε, πιστεύω τελικά ότι μετά από τις συζητήσεις θα ε, συζητήσουμε και θα καταλήξουμε σε μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, ίσω αυτή ήταν η καλύτερη ομιλία που έκανα ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα ωραία μας τα λέτε. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η καλύτερη. Εν πάση περιπτώσει. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο Άλφερτ Σάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, συνεργασία και την πρόθεσή του να βρούμε συμβασμούς επί του κειμένου. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να περιοριστούμε σε μία προσέγγιση με βάση τις αρχές, τις βέλτιστες πρακτικές και τα εθνικά συστήματα που όπω έχουμε πολλές φορές λειτουργούν πολύ καλά μέχρι τώρα και δεν θα πρέπει εμείς να του δημιουργήσουμε προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίε, εμείς έχουμε υποβάλει ε, πάνω από 70 ε, τροπολογίε για την οδηγία για τον κανονισμό. Όπως είχε πει ο εισηγητή και κατά το παρελθόν, ε, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το κείμενο τη οδηγία μεταξύ σκιωδών. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και επειδή η ψηφοφορία ε, θα γίνει σε δύο εβδομάδε, πρέπει να επιταχύνουμε. Τα βασικά στοιχεία για μα έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του εισηγητή στα εξή ζητήματα. Επιλέξουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται ε, κανονικέ κανονικές ομολογίε ομολογίες ε, ή συνήθεις, συνήθους Ε, πάμε στοιχεία πρέπει να παραμείνουν στο κείμενο και τρίτον στη σύνθεση της κάλυψης ε, της ομάδας που είναι ιδιαίτερα περιοριστική. Στα άρθρα 11 και 15 πρέπει να σταθούμε σε συνδυασμό με τη συζήτηση για τον κανονισμό CRR. Εδώ πέρα βέβαια δεν έχουμε ακόμα εξετάσει την πρόταση αναθεώρησης του CRR. Το άρθρο όμω 129 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και θα έχει άμεσε επιπτώσει και σε άλλου τομεί. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την προτιμησιακή ε, αντιμετώπιση, ε, στην τροπολογία 14 αναφέρεται προηγουμένως ε, και το soft bullet, θα δοθεί έτσι ένα ασφαλμένο μήνυμα προς τους επενδυτές. Για να εξομαλυνθεί η διαδικασία όμως πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σαφές το κείμενο. Ε, να σταθούμε μόνο σε αυτά που έχουν αξιολογηθεί αντικειμενικά και να αποφύγουμε ε, αναταραχές στις αγορές. Ευχαριστώ. Καρολίνη Ταγκάλ από την Άλντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο καλυμμένων ομολογιών στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής της Ένωσης Κεφαλαγορών. Έχουμε μια τέτοια πρόταση που θα μας δώσει μια σταθερή και προστατευμένη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές. Και το προτινόμενο πλαίσιο δίνει ε, δυνατότητες ασφαλών επενδύσεων και μεγαλύτερη ε, οικονομική σταθερότητα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, στηρίζουμε τη φύση τη ε, πρόταση οδηγία, καθώ επιτρέπει ε, σε επιτρέπει ελάχιστη εναρμόνιση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε τα υψηλότερα δυνατά ε, πρότυπα για τις καλυμμένες ομολογίες και να αποφύγουμε τα χαμηλής ποιότητας. Εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογίες στο άρθρο 6 που περιορίζουν το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας ε, στις ε, καλυμμένες οδηγίες που τηρούν τις κοινέ κανονικές κεφαλαϊκές απαιτήσει. Η πρόταση του κυρίου Λούκε μπορεί να αποτελέσει καλή βάση συμβασμού για όλους μας. Φυσικά πρέπει να οριστικοποιήσουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα για τις καλυμμένες ομολογίες. Να πω ότι ήδη έχουμε μιλήσει για την ε, παράταση στην ορίμανση και σε προηγούμενες συνεδριάσεις και να επισημάνω ότι ε, οι εξολογήσει υψηλού κινδύνου για συγκεκριμένε ομολογίε ε, είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ, αλλά το ξέρετε αυτό. Γιατί ε, δεν στερίζεται και από στοιχεία που προκύπτουν από την αγορά. Θέλω λοιπόν να τα συζητήσουμε περαιτέρω αυτά στους συντονιστές και να εγκριθεί σύντομα η έκθεση για να υπάρξει συμφωνία σε πλαίσιο τριμερούς διαλόγου ε, πριν το τέλος της θητείας. Ελπίζω αυτό να καταστεί εφικτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από τους πράσινους ο κ. Λάμπερτς. Ε, όντως, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Λυπάμαι κύριε Σιγητά που δεν ήμουν και πολύ παρόν μέχρι στιγμή στην όλη διαδικασία. Πάντως εκτιμούμε ε, τις πρώτες εξελίξεις ε, των αρχικών συμβαστικών τροπολογιών. Έχουμε έχετε λάβει υπόψη αρκετές ανησυχίες μας, κύριε Σιγητά, και σας ευχαριστούμε, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ακόμη κάποια θέματα. Έχουμε τέσσερα προβλήματα με τις συμβαστικές τροπολογίες. Επιτρέπουν αντί να απαιτούν την, το διορισμό ενός επόπτη καλυμμένων ομολόγων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτικό αυτό το μέτρο. Επίσης, δεν ζητά δημοσιοποίηση επιπλέον πληροφοριών για διάφορα καλυμμένα τέτοια ομόλογα, ακόμη και για στεγαστικά ενυποθεκά δάνεια και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία. Επιτρέπει τη συμπερίληψη λιγότερο ρευστών στοιχείων όπως ομόλογα εταιριών ή τιτλοποιημένα ομόλογα στο, στη δικλίδα ασφαλείας για τη ρευστοποίηση και προβλέπει διοικητικά μέσα για προσφυγές σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας. Ό,τι αφορά τον κανονισμό, ε, δεν, δεν έχουμε λάβει ακόμα τις συμβαστικές προτάσεις ή τις βασικές τροπολογίες ε, για να υιοθετηθεί υψηλή ποσότητα των ε, καλυμμένων ομολόγων, περιορίζοντας το άνοιγμα σε χρηματοπιστωτικά ίδρυμα που, θεωρώ, που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία ναι. και επίσης θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές ε, για τα επιλέξιμα αυτά περιουσιακά στοιχεία. Ε, ζητούμε ε, ελάχιστα επίπεδα με βάση τις συνθήκες της, της Σύμβασης Βασιλείας και η απέτηση για υποκατάστατα ομόλογα θα πρέπει να θεωρούνται ως ποσοτικός περιορισμός. Αυτά, αυτά είναι ο προβληματισμός μας και περιμένουμε συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Θέλουμε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτική θητείας ε, να ολοκληρώσουμε, να διεκπαιρώσουμε αυτό το θέμα. Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά επειδή είναι και πολύ περίπλοκο, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Um, and... Uh, σας ευχαριστούμε. Πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ δεν βλέπω, ούτε ΕΝΦ, η FTD. Yes, but First, we have the catch the eye, and then we go to the commission. So, um, for catch the eye... Επιτροπή, catch the eye. Δεν βλέπω να στάει κανείς. Ε, αντάς πω και εγώ δύο λόγια. Εν γέννη λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στο στόχο ε, της υιοθέτηση αυτού του ε, νομοθετήματος. Στόχο θετικό, Λαμβανωμένη υπόψη τη σημασία των καλυμμένων ομολόγων και τη ανάγκη για μια καλή εξισορρόπηση, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, δηλαδή αφενός με να υπάρξει εναρμόνιση της αγοράς, ταυτόχρονα όμω, και να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο προϋποθέσεων εναρμόνισης για να γίνονται σεβαστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υφισταμένων αγορών αλλά και η ανάγκη της προστασίας του καταναλωτή και της δημοσιονομικής σταθερο... δι... χρηματοπιστωτικής νομής σταθερότητας. Επίσης, σε κάποια σημεία που βλέπουμε ότι ορισμένες τροπολογίες ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, καταρχάς τα εισπαράγωγες συμβάσεις σε προγράμματα καλυμμένων ομολόγων. Και αν συνδυάσουμε τα άρθρα 11 της οδηγίας και 129 της οδηγίας ε, CRR που μας λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έτσι περιορίζονται οι ε, επιλέξιμοι φορείς σε αυτούς μόνο που έχουν αξιολόγηση ποιότητας 1 και 2, άρα περιορίζεται αρκετά το πεδίο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θεωρούνται ε, ικανά για επένδυση και ταυτόχρονα θα ανεβάσει την πίεση σε τράπεζες ε, χαμηλότερης ε, αξιολόγησης σε ορισμένες χώρες με συνέπειες ενδεχομένως και τη συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση των αγορών και του ενεργητικού που θα θεωρηθούν ως πρώτης και δεύτερης βαθμίδας από τις αγορές. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτός ο περιορισμός δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητες μέθοδοι για την αξιολόγηση της ε, ποιότητας των ε, αντισυμβαλωμένων και αρκούν αυτοί. Επίσης, άρθρο 16 δύο περιορισμένες κατηγορίες για την αξιολόγηση του ενεργητικού ρευστότητας ε, για οργανισμούς δεύτερης και τρίτης βαθμίδας. Τροπολογίες καλές πιστεύω. που εξασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση για, όλ, για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλων των βαθμίδων αλλά με διαφορετικές κατευθύνσεις κάθε φορά και έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα τρόπο τον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται παραδείγματι με κάποιες ε, διασφαλιστικές σε σχέση με την, ε, ανάλογα με την βαθμίδα και χάρη στην στήριξη των εθνικών αρχών. Αυτό, αλλά πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα παρακαλέσω την Επιτροπή Ευχαριστώ. And, uh, for... Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλου του ομιλητέ. Ήταν καλό η βάση συζήτηση στο σχέδιο και οι τροπολογίε νομίζω θα μπορέσουν να βρουν τη θέση του μέσα στην έκθεση. Πολλέ έχουν να κάνουν με τη συνέπεια σε ήδη λειτουργούσε σε εθνικέ αγορέ με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου και δεν διαταράσουν, δεν φαίνεται να διαταράσουν τι εθνικέ αγορέ. Ε, Επίσης είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τη σταθερότητα των αγορών ε, όταν κάνουμε τη ρύθμιση των καλυμμένων ομολόγων. Είπε και ο εισηγητής ότι έχουμε σημεία σημαντικά στα άρθρα 6, 6α που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και δι. στο πόσο θα πρέπει η πίεση εποπτική να αυξηθεί και ενδεχομένω να επεκταθεί και σε άλλο ενεργετικό πέραν των καλυμμένων ομολόγων ε, με διαφορετικές τεχνικές. Πάντως πολύ καλή πρόταση και συγχαρητήρια στο Κοινοβούλιο που προχώρησε τόσο γρήγορα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια. Τους ε, σκιώδη ηγητές, τους συναδέλφους, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα που εξακολουθεί να παραμένει επίμαχο. Την αντιμετώπιση της ε, στάθμης κινδύνου για, κάποι, για την παράταση της λικτότητας. Ε, θα ήθελα να θεωρήσετε την αρνητική σας στάση απέναντι στην πρότασή μου για, την, για το θέμα αυτό της παράτασης λικτότητας και πώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη στάθμιση κινδύνου. Οι παρατηταμένες ε, λικτότητες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί βάθος. Ούτε το θέμα της στάθμισης ε, κινδύνου έχει εξεταστεί αναλυτικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα των ε, επεκτηνόμενων αλεκτοτήτων ε, δεν έχει αναλυθεί ούτε από την Κεντρική Τράπεζα, ούτε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συστηματικά. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασαν ανησυχίε για τέτοιου είδου δομέ. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι το, η έκθεση της Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών του 2016 αποσαφηνίζει ότι κατά τη γνώμη τους αυτές οι επικριταμένες λεκτότητες ε, δημιουργεί προβλήματα στον επενδυτή και από άποψη υποπτίας και από άποψη κανονιστικής ρυθμίσης. Οπότε και από άποψη συμφωνίας της Βασιλείας και μακροληπτικού κινδύνου, γιατί μπορεί να είναι επιτυχή στην αγορά, αλλά δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε περίοδο κρίσης και δεν ξέρουμε τι κίνδυνοι ρευστότητα θα πρέπει να αναλάβουν οι επενδυτέ σε περίπτωση που έχουν καλυμμένα ομόλογα με παρατεταμένη ληκτότητα. Επίσης, αυτή η ιδέα της παράτες λεκτότητα παραβιάζει την αρχή της διπλής προσφυγής, που είναι ε, βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας του εκδότη. Με αυτά τα σχόλια λοιπόν θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον Πρόεδρο, ευχαριστώντα και πάλι τους συναδέλφους για τα επικοδομητικά του σχόλια και προσβλέποντας τη συνέχιση των συζητήσεων. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους συναδέλφους και την Επιτροπή. Θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ 5 Νοεμβρίου. Οπότε φροντίστε να βρείτε συμβαστικές τροπολογίες καιρός, για να προλάβουν να ψηφίσουμε στην προγραμματισμένη ημερομηνία ώστε να περάσει την πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου το θέμα. Ευχαριστώ. Σε έξι λεπτά θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Colleagues, uh, please take seat. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη.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 Ξεκινούμε λοιπόν με τα αποτελέσματα των ε, διοργανικών διαπραγματεύσεων για την έδρα της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρας. 36 υπέρ, 4 κατά, 0 εποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που πλέον έχει και έδρα. Ας περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Μαυρίδη, οικονομικές πολιτικές στην Ευρωζώνη, συμβαστική γάμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται νομίζω, αλλά την ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 18 κατά. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική E. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ κατά ελέγχουμε τη σημαστική F. Πέρας. Απορρίπτεται 19 κατά 16 υπέρ. Πάμε λοιπόν στις, στην ε, τροπολογία 79 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 79 άρχεται η Και ο εισηγητή, αν βιαστεί μπορεί και να ψηφίσει. Σύντομα παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, 2 αποχές. Εάν εγκριθεί, λέει, εγκ... καταπίπτουν οι υπόλοιπες. Πάμε λοιπόν στην 91 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Συμβαστική H. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε? Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική H, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 23 ψήφοι κατά, 17 υπέρ. Πάμε λοιπόν. Το 10 και το 11. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε τη 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Γιατί είναι μικρή η διαφορά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέρας. Και πάλι 20 κατά 19 υπέρ. Απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 102. Αρχίτε. Ένας μένει ακόμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 κατά, 17 υπέρ. 103 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 103. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 κατά, 19 υπέρ. 104 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε και την 104. Πέρας, απορρίπτεται. 20 κατά, 19 υπέρ. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 106. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 16 υπέρ. 107 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 107. Πέρας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι για την 108. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 19 κατά. Μπορούμε να ψηφίσουμε και την 109. Δεν έχω καταλάβει αν καταπίπτει. Ωραία, ψηφίζουμε για την 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε του αρχικού κειμένου. Ας περάσουμε στην 110. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112. Υπέρ, κατά. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 113. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική I υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την 138 τροπολογία υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 140. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 141. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ 18 κατά. 146 κατά πίπτη. Ας ψηφίσουμε την 142. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 142. Πέρας. Έγκρινεται. 143. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 143. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146. Α, όχι. Την 147 πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 147. Απορρίπτεται. Καταπίπτει και η ψήφος για το αρχικό κείμενο. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 149 Πέρας. Έγκρινεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά ελέγχουμε την 152 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ισοψηφία επομένω απορρίπτεται 153 υπέρ κατά ελέγχουμε την 153 Πέρας. Και πάλι ψηφία Απορρίπτεται. 154. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 19 κατά. 155 υπέρ. Κατά ελέγχουμε και την 155. Πέρας. Απορρίπτεται. 156. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 156. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ομικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την Q. Vote is closed. Πέρας. Απεριφθεί. 20 υπέρ, 23 κατά. 203 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 204 υπέρ, κατά. Και επαληθεύουμε. 204. Πέρας. Απορρίφθηκε. 20 κατά 19 υπέρ. 205 υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε παρακαλώ. One vote. Ακόμα ένας πρέπει να ψηφίσει. Πέρας. Απεριφθεί με 20 ψήφους κατά. 206 υπέρ. Επαληθεύουμε. Πέρας. Ε, η ψηφοφορία παρακαλώ. Και πέρας. Ισοψηφία και περίφθη 207 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. 207. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία και πάλι απερίφθη. 208 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε τη 208, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Με 21 ψήφους κατά. 209 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη. 210 υπέρ. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Πέρας. Ισοψηφία και περίφθη. 211 υπέρ και επαληθεύουμε. Πέρας. Ισοψηφία και πάλι απερίφθη. 212. Υπέρ. Επαληθεύουμε τη 212. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Adopted 24 in Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Δεν ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο λοιπόν και πάμε στη 213 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 214 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 217 υπέρ κατά και επαληθεύουμε. Vote is closed. Πέρας. Και ισοψηφία με απόρριψη. 218 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές απερίφθη. 219 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 220 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 221 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 222 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 223 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 215 υπέρ κατά επαληθεύω, 215 πέρας και απερίφθη. Συμβαστική R, ρο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική S, σίγμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. T, ταφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική U, υπέρ, κατά, υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την U, συμβαστική U. Πέρας και εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ, 19 κατά. Συμβαστική Β, Β, υπέρ, κατά, υπέρ, κατά. Αποχές και εγκρίνεται νομίζω, αλλά σε επαληθεύσουμε αν θέλετε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και δεν εγκρίθηκε. Α, οι φιλελεύθεροι που πριν ψήφισαν υπέρ τώρα καταψήφισαν. Ναι, αλλά Α, αυτό ήτανε. Καλό ήτανε που επαλήθευσα. Νομίζω ότι είχαν υπερψηφίσει και οι φιλελεύθεροι, αυτό θεώρησα πως έχει εγκριθεί. Ωραία, τότε πάω στην 2.90 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Με 21 ψήφους κατά. Η 291 ήταν ταυτόσιμοι τους ή άλλως. 292 υπέρ κατά. Καλά επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με 21 ψήφους κατά και 20 υπέρ. 293 υπέρ. Επαληθεύουμε. 293. Πέρας και απερίφθη με 23 ψήφους κατά και 20 υπέρ. 294 υπέρ. Επαληθεύουμε. Πέρας και απερίφθη 25 ψήφους κατά και 18 υπέρ, 295 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. 23 ψήφοι κατά, 20 υπέρ, 296 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. 23 υπέρ, 19 κατά. Παράξερο να υιοθετείτε το αρχικό κείμενο ενώ έχει απορριφθεί η συμβαστική τροπολογία. 297 υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε. Απε... Α... Άρχεται ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. πέρασε ψηφοφορία Και απερίφθη. Με 23 ψήφους ε, κατά 19 υπέρ. 298 υπέρ. Και επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραν της, πέρας της ψηφοφορίας με 21 ψήφους κατά 299. Ας επαληθεύσουμε κατευθείαν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Vote is closed. Rejected. Απερίφθη. 300 ηλεκτρονικά κατευθείαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed πέρας και απερίφθη. 301 αρχίζουμε ηλεκτρονικά. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο δεν μπορούν να μεταφραστούν. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απερίφθη συμβαστική W υπέρ. Και παρακαλώ να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 22 υπέρ 19 κατά. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Y y υπέρ και επαληθεύουμε. Πέρας. Ισοτιμία και ε, ισοψηφία και απερίφθη 319 υπέρ. Επαληθεύουμε παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. πέρας και απερίφθη. 320 ήταν ταυτόσημη, 321 τώρα. Α, όχι. Στην 300 και η 321 ταυτόσημη, 322 τώρα, υπέρ. 3, 2, 2 και επαληθεύουμε. Πέρασε απερίφθη. 323 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 324 υπέρ κατά και επαληθεύουμε. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. ψηφία και απερίφθη αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Το κλείσατε πολύ γρήγορα το σύστημα. Ε, ξαναρχίζουμε την ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Αρχικό κείμενο. Έχουν μείνει κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Στην επανάληψη παρακαλώ. Και πέρας. Ισοψηφία και απερίφθη. 325 υπέρ και επαληθεύουμε. Πέρας και εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 326 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Πέρας απερίφθη 327 υπέρ και επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη με 20 ψήφους κατά και 20 υπέρ, 328 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη. Συμβαστική A, α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β, υπέρ και επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη με 21 ψήφους κατά. Τροπολογία 3 τότε υπέρ και επαληθεύουμε. Πέρας εγκρίνεται. Και άρα ψηφίζουμε και την 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 24 υπέρ κατά. Και επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Με 23 ψήφους κατά και 18 υπέρ. 25 υπέρ. Επαληθεύουμε. Την 25 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με 21 ψήφους υπέρ και 19 κατά, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 28 υπέρ κατά και επαληθεύουμε την 28, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη με 20 ψήφους κατά και 19 υπέρ, 29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 30 επαληθεύουμε την 29. Πέρας. 15 υπέρ, 24 κατά και απερίφθη, 30 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη 31 υπέρ. Και επαληθεύουμε την 31. Πέρας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, κατά και, ε, υπέρ και 18 κατά. Και άρα πάω στην 30, όχι, 32 ε, υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 32. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και 19 κατά. 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 34 υπέρ. Επαληθεύουμε την 34 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη 35 υπέρ κατά επαληθεύουμε την 35 πέρας απερίφθη 36 υπέρ και επαληθεύουμε την 36 πέρας απερίφθη 37 υπέρ κατά Επαληθεύουμε την 37. Πέρας. Απερίφθη. Με 20 ψήφους κατά. 38 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Ισοψηφία και απερίφθη 39 υπέρ. Επαληθεύουμε. Α, εγκρίνεται. Πέρες προφορίες, εντάξει, είναι σαφές ότι εγκρίθηκε, ε, συγγνώμη για το λάθος, 40 υπέρ, κατά και επαληθεύω. Πέρας απερίφθη. 23 ψήφι κατά 16 υπέρ, 41 υπέρ κατά και επαληθεύουμε. Περ, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους κατά 19 υπέρ, 42 κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ κατά επαληθεύουμε παρακαλώ πέρας και απερίφθη 45 υπέρ 45 υπέρ κατά επαληθεύουμε τις 45 παρακαλώ Πέρας. Απερίφθη με 21 ψήφους κατά και 20 υπέρ. 46 υπέρ. Ελέγχουμε. Πέρας. Απερίφθη 21 ψήφους κατά 20 υπέρ. 47 υπέρ. Επαληθεύουμε. Πέρας. Ισοψηφία και απερίφθη υπέρ 20 κατά. Ε, μετά έχουμε τροπολογία υπερθυμών 1 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 1. Πέρας. Απερίφθη 2 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε και τη 2. και εγκρίνεται 4 υπερκατάποχες αποχές απερίφθη 9 υπερκατάποχες αποχές απερίφθη 266 υπερκατάποχες αποχές απερίφθη 267 υπερκατά επαληθεύουμε τη 267 Πέρας. Απερίφθη 24 κατά 20 υπέρ. Και τώρα, κατόπιν ετοίματος των ομάδων, θα κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή για να γίνει ανάλυση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, που είναι τόσο περίπλοκη, με πολλές συμβαστικές που απερίφθησαν. Uh, Συνάδελφοι, επιστρέφουμε στην ψηφοφορία. Paradoxically, produce less incoherence that one might. Τελικά δεν υπάρχει τέτοια ασυνέπεια που περιμέναμε μετά από τόσες πολλές ψηφοφορίες η ασυναρτησία μάλλον. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Still two colleagues to vote. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Vote is closed. against 20. Απορρίπτεται με 20 ψήφους υπέρ και 22 κατά ο κύριος Βανκέντελα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Λυπάμαι, λυπάμαι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σήμερα. Γιατί δεν ε, καλή εντύπωση που δίνουμε όταν δεν καταφέρνουμε να εγκρίνουμε τόσο σημαντική έκθεση. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίες είχαμε στενή συνεργασία με τον εισηγητή και επικοδομητική και ελπίζω εν ώψη της Ολομέλειας να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις. Ο εισηγητής θέλει να πει κάτι. I be quite short. Um, I appreciate... Μάλιστα, εν συντομία. Εκτιμώ αυτό που είπε ο συνάδελφο, θα συζητήσουμε περαιτέρω αλλά απ' την άλλη για μας ε, είναι απογοητευτικό το γεγονό ότι... Γιατί τελικά αυτή η έκθεση έχει πολύ περισσότερες προεκτάσεις από τα όσα συζητήθηκαν για το ίδιο το έγγραφο. Απευθύνω έκκληση προς όλους όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται ε, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να το ξανασκεφτούν. Αυτό ήθελα να πω μόνο προς όλους στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Θα δούμε ποια θα είναι διαδικαστικά τα βήματα από εδώ και πέρα. Πάντως ε, είναι αρνητικό το ότι απορρίφθηκε η έκθεση. Θα σε ενημερώσουμε πάντως για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα διαδικαστικά. Περνάμε παρακαλώ ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί για την έκθεση αυτή που δεν είναι έκθεση αλλά γνωμοδότηση, ε, θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Οπότε ε, θα δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Ίσως θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την ε, αρμόδια κατουσία Επιτροπή που είναι η Γιούρη. Και ελπίζω στο μεταξύ εκκρεμότητες να διαθετηθούν και φαντάζομαι ο εισηγητή και οι σκιώδει εισηγητέ θα θελήσουν να επηρεάσουν κάπως το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης τη επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ναι, ναι, αλλά μιλάμε για το νέο κείμενο που θα ψηφίσουμε. Υπερβάνς. Καταλαβαίνω αυτό που υπονοεί ο Αντρέας Φαπ, γιατί το ΕΛΚ τελευταία στιγμή έβαλε ε, ψηφοφορία κλειδί key vote για μια συμβαστική πρόταση για να ε, ε, ε, εξαιρέσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από την ιδεολογική σκέψη F. Αν τελικά περάσει, έπρεπε να δώσουμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νορικών Υποθέσεων, Νομικών Υποθέσεων. Οπότε αυτοί που ήταν κατά αυτή τη key vote θα μπορούσαν να κερδίσουν το χαμένο έδαφο και να επανέλθουν στην Νομική Επιτροπή. Να σα πω περί τίνο πρόκειται γιατί εδώ όλοι έχουμε δεσμευθεί να είμαστε ανένδοτοι με βάση και την επικαιρότητα, να είμαστε ανένδοτοι στην καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ ε, απαλλάσσουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από το μηχανισμό και τις ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπουμε για τις επιχειρήσεις που κάνουν συγχωνεύσεις ή διασπάσεις. Ενώ γνωρίζουμε ότι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να κρύβονται άλλες επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, επιχειρήσεις προπετάσματα. Ε, οπότε προσοχή ε, τι θα ψηφίσουμε. Γιατί για το ΕΛΚ είναι key vote, αλλά και για μας το ίδιο. Ας απομιστούμε λοιπόν τις ευθύνες μας και να μην υπερψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σβάμπ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία Α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 195. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σ, Α, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία CA. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 21 προς 20. Τροπολογία 206. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 206. Άρχεται η ψηφοφορία. 206. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Ι. ε με προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σβάμπ. Ψηφίζουμε. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Αν θέλετε έλεγχο, ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε στη συμβαστική τροπολογία ε. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική ε. Περβάς, προτείνεις κατά. Yeah, okay. Good. Μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F με την προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σβάπ και πάλι. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον έχει απορριφθεί όμως. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Με 24 ψήφους υπέρ, και 19 κατά. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία G. Ποιος είναι υπέρ. G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 276. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 276. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 προς 19. 277. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 277. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 21 ψήφι υπέρ, 20 κατά, 2,78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 2,79 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 279 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 21 προς 20. 280. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 281. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 286 άρχιτη ψηφοφορία Τέλος. Απορρίπτεται. 19 προς 23. H. Συμβαστική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 289. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 289. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 20 προς 22. 290. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.91 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.91 άρχεται η ψηφοφορία Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 20 προς 22 2.92 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 2.92 άρχεται η ψηφοφορία τέλος Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 2.93 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.93. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Τέλος. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 2.94. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 2.94. Θα έλεγα ότι μάλλον ε, εγκρίνεται, αλλά είναι οριακό το αποτέλεσμα. Ισοψηφία απορρίπτεται. 2,90, όχι το 2,95 είναι γλωσσικού χαρακτήρα. 2,95, πρέπει και αυτό να το ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 295, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 296 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 296. Τέλος. Ισοψηφία και πάλι απορρίπτεται. 2,97. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2,97. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 20 προς 21. Συμβαστική τροπολογία I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 προς 19, 19 προς 21. 328 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 328. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. ισοψηφία απορρίπτεται. 329. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 329, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 330. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 331 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη υπέρ με την προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σφάπ. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία π υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q υπέρ κατά Κατά εγκρίνεται. 347 τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 348 υπέρ. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ρο, υπέρ, αρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S, με την προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σβάπ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε την, συμβαστική τροπολογία χωρίς την προφορική του ΣΒΑΠ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 365. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές, μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε καλό κακό, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΤΑΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 374 υπέρ κατά αποχές, α μάλλον 374 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται, 375 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται, 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 378 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 380 άρχεται ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται με ισοψηφία τροπολογία 90 υπέρ κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 20 προς 22 απορρίπτεται. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 382 της ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 22 προς 18. Συμβαστική τροπολογία V υπέρ κατά αποχές ε, ε, συγγνώμη, V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 390 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για 390 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται 20 προς 22. 391. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιο υπέρ, συγγνώμη, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ισοψηφία και πάλι απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία W. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία YA υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία YA. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται 20 προς 21. Εναλλακτική YA υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την εναλλακτική YA άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 22 προς 19 συμβαστική τροπολογία Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 413 υπέρ υπέρ 413 κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία αα με προφορική τροπολογία του Ανδρέα Σφάπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε ή μάλλον Ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία ΑΑ, τη συμβαστική. Χωρίς την προφορική το κύριο Σβάπ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΒ. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AC. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 451. 451. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 452. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 453. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 454. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 455 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 456 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 457 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 458 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 459 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 460 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 461 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική τροπολογία AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 464 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 465 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AF συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 485 υπέρ κατά. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 485. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 20 προς 19. 486. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AHA υπέρ κατά αποχές με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 98 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται 100 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 100 άρχιτη ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 20 προς 19 101 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχιτη ψηφοφορία Τέλος, εγκρίνεται. 20 προς 19. 102 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 102. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 20 προς 19. Συμβαστική τροπολογία ΑΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 105. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, ισοψηφία απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική αλφα λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 110. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 προς 19. Συμβαστική τροπολογία αλφαμή υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 113 η ψηφοφορία. Τέλος. Ισοπαλία και πάλι 20... Οπότε απορρίπτεται 114 υπέρ κατά απορρίπτεται, τροπολογία 7 υπέρ, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 7, άρχεται ψηφοφορία. Vote Τέλος. 2020 Η ισοψηφία απορρίπτεται. 115 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is Τέλος. Εγκρίνεται 20 προς 19. Συμβαστική τροπολογία αλφανή. Ναι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται αλφα όμικρον. Υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Ομικρον συμβαστική άρχιτη ψηφοφορία. Is closed. Τέλος. So... Απορρίπτεται. 129, 129 συγγνώμη, άρχιτη ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Rejected απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 122 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Να ελέγξουμε την 123 άρχεται. Πέρα. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Ας ελέγξουμε την 125. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ. Ας ελέγξουμε για τον 126. Πέρας. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Ελέγχουμε για την 127. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 129 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Ελέγχουμε την 131. Πέρας. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Ελέγχουμε. Άρχεται η Ολόκληρο βιβλίο έχουμε γράψει, Σβέν. Γεμάτα τελογικές σκέψεις. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική AP, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AQ, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 138, πίπτη, συγγνώμη. Συμβαστική AR, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 142, υπέρ Ας ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Ελέγχουμε την 145. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Ελέγχουμε την 148. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 150 Πέρας. Εγκρίνεται. 151. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές α... Ταυτόσιμες δύο τροπολογίες του ίδιου, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τέλος πάντων, απορρίπτεται επανάληψη μη τριμαθήσεως λέμε. Ωραία, 155 υπέρ. Κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Συμβαστική AS, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ, ελέγχουμε την 161 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 162. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 163. Περ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 165. Vote is closed. Πέρας. Έγκρινεται. 166 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τον 166. Vote is closed. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τον 167. Vote is closed. Πέρας. Ισοψηφία. Έφυγε ένα πράσινο, χάνοντα την πλειοψηφία. Ε, συμβαστική AT υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 173 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 173. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 194 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 195. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 179. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AU. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 187 ελέγχουμε. Προβλέψουμε πλέον κατάσταση. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Α, τα ψηφίσαμε αυτά. 188 απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Για την πρόταση τώρα της... Α, συγγνώμη, θέλετε διάλειμμα. Μάλιστα. Alex, take seat, please. Καθίστε παρακαλώ. Vote now. Καθίστε για να ψηφίσουμε. Καθίσατε όλοι, είστε έτοιμοι. Ωραία. Να ψηφίσουμε επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει τροποποιηθεί. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 36 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές. Έγκρινεται η νομοδότηση. Συγχαρητήρια. Please. Σβέν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε σημαντική καθυστέρηση στις ε, διεργασίες της Επιτροπής, στο τέλος της μέσης διάταξης έχουμε την έκθεση του ανταγωνισμού. Επειδή ο εισηγητής είναι από τους πρασίνους. Θα μπορούσε να μετατεθεί για άλλη συνεδρίαση η εξέταση της έκθεσης για να διευκολύνουν την κατάσταση σήμερα. Είναι και ένα μικρό δώρο προς τη διερμηνία και προς ε, τους σκιώδεις. So now we go on with the agenda. We try... Ωραία, συνεχίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έχουμε εδώ... και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι πολύ αυστηρός ό,τι αφορά τον ε, χρόνο μιλία. Σας το λέω από τώρα. Πολύ πολύ αυστηρός. Λοιπόν, σημείο 9 η έκθεση της κυρίας Νίνα Γκίλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ξέρω ότι ήταν μακροσκελής ε, η διαδικασία των ψηφοφοριών. Παρακαλώ, ησυχία. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές επενδυτικές προκλήσεις, ε, σε ό,τι αφορά την ε, εκπλήρωση των στόχων για το περιβάλλον μέχρι το 2030 χρειαζόμαστε κάθε χρόνο επιπρόσθετη χρηματοδότηση 180 δισεκατομμυρίων στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος μόνο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από το δημόσιο τομέα. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικές προσπάθειες και από τον ιδιωτικό κλάδο. Γι' αυτό ε, και χαιρετίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα ω ένα βήμα προς ε, πιο βιώσιμο χρηματοοικονομικό σύστημα. Σημειώνω επίση τι προσπάθειε ε, που καταβάλλονται από του παρόχου δικτών ε, για την ε, ανάπτυξη μεγάλου φάσματος δικτών που θα λαμβάνουν υπόψη και τους στόχους της βιωσιμότητας και του κλίματος. Ο ο τομέα των δικτών αναφορά έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και συμφωνώ με την εκτίμηση ότι οι ε, χρηματοοικονομικοί δείκτε αναφορά είναι ακραγωνιαίο λήθο ε, των χρηματαγορών και πολλοί επενδυτέ ε, βασίζονται στου δείκτε αναφορά για να μετρήσουν την απόδοση συγκεκριμένων προϊόντων και για να κατανείμουν τα χρηματοφυλακιά του. Όμω υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με, το, το σύνολο της οικονομίας, γιατί μόλις με 10,3% των ε, ε, χρηματοοικονομικών ε, δικτών αναφοράς έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση σήμερα. Συμμερίζομαι και τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει η ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς ως βασικό κινητήριο μοχλό μιας βραχυπρόθεσμης προσέγγισης που δεν συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και έτσι συμβάλλουμε περισσότερο και κατευθυνόμαστε κατευθυνόμεθα προ την κατανομή χαρτοφυλακίων που δεν συνάδουν με του μακροπρόθεσμου στόχου ε, βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Αυτά είναι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε με αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ε, να παρέμβουμε εδώ ως ε, νομοθέτες με βάση και με την έκθεση της πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για την βιώσιμη χρηματοδότηση πρέπει να επιδείξουμε ρεαλισμό, ανοιχτό πνεύμα και να ακολουθήσουμε την καινοτομία. Είναι σημαντικό ταυτόχρονα να δώσουμε και στον κλάδο ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια ό,τι αφορά την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε. Θεωρώ ότι ο στόχος πολιτικής είναι σαφός. Ε, πρέπει να πετύχουμε τους στόχους πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί από εμάς και να επιδείξουμε τα επίπεδα φιλοδοξίας που προκύπτουν και από άλλα τμήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να εφαρμόσουμε, να ελοποιήσουμε ε, τα στοιχεία αυτά, ε, σύστημα ITS, νομοθεσία περικτηρίων και το καθεξής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει... Ε, δεν υπάρχουν παρανοήσεις, προς τους επενδυτές αυτό που λέγεται greenwashing, δηλαδή ε, ένας ψευδοπράσινος ε, χαρακτήρας. Πρέπει λοιπόν, και αντιτίθεμαι στην ιδέα ότι, ή μάλλον συμφωνώ με την, με την έννοια ότι πρέπει να εντάξουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας σε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Γι' αυτό έχω θέσει και την προθεσμία του 2022, τόσο ώστε οι πάροχοι δικτών αναφοράς να μπορούν να δημοσιεύσουν ε, τους δείκτες αναφοράς που συνάδουν με τη Συμφωνία των Παρισίων και σε σχέση με ζητήματα που έχουν υλοποιηθεί σε άλλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πρέπει να τυποποιήσουμε τη μεθοδολογία και αυτό να γίνει μέσω κατεξοδότηση πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα δημοσιευθεί εντός διετίας από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού. Για τους επενδυτές απαραίτητο είναι να έχουν σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες και γι' αυτό θέλω να υπάρχει περιγραφή κατά τρόπο ακριβή και τυποποιημένο των οροσίμων από αυτούς που τα ορίζουν και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τα ορόσημα αυτά κινούνται και τον τρόπο με τον οποίο προς τις ε, προς τη Συμφωνία των Παρισίων. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται κάπως παρεμβατικό, ριζοσπαστικό. Δεν υπάρχουν όμως επαρκώς επιλέξιμα ε, προϊόντα που να πληρούν. Δέκα δευτερόλεπτα, Ρίνα, που να πληρούν τα κριτήρια. Δέκα δεύτερα. Καλά, να κλείσω λοιπόν. Διαφωνώ λοιπόν με αυτό το επιχείρημα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τομεί που μεταλλάσσονται ταχύτατα και μπορούμε στο μέλλον να δούμε καλά αποτελέσματα. Πρόεδρε, αν έχετε την ευκαιρία άλλη φορά να μου δώσετε το λόγο. Αν σαντέχ, τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις που μας έχει κάνει. Κάποιοι από τους τομείς ήδη έχουν ε, αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείμενο ενδιαφέροντος για ένα πρασίνισμα της οικονομίας. Τώρα πρέπει πια να κινηθούμε και προς το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, οι πράσινοι δείκτες λοιπόν έχουν κινηθεί αρκετά, χωρίς όμως ένα πραγματικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Τώρα γιατί μπορούν να δώσουν ε, ακριβή και αξιόπιστη εικόνα της, ε, του οικονομικού περιβάλλοντος. Για να μπορούν να δώσουν λοιπόν ακριβή εικόνα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μία προσέγγιση με βάση δύο δείκτες, ε, είτε χωρίς άνθρακα είτε θετικό ε, ισοζύγιο άνθρακα, που μπορούν να είναι σαφείς και να προσελκύσουν τους επενδυτές. Τους ορισμούς ίσως χρειαστεί περισσότερη σαφήνεια για να μην ε, ξεγελάμε τον καταναλωτή με το greenwashing. Για τις προτάσεις της εισηγήτριας. Έως το 2022 μας προτείνει όπως μας είπε, όλοι αυτοί οι δείκτες να μετατραπούν σε θετικού ισοζυγίου ως προς τον άνθρακα. Μου φαίνεται υπερβολικά ριζική και δύσκολα εφαρμόσιμη η πρότασή της όμως. Όντως, ο αριθμό των επιχειρήσεων που θα ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία των Παρισίων, με τις Συμφωνίες των Παρισίων βεβαίως θα αυξηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένο ο αριθμό του. Επομένως, πώς μπορούμε να χτίσουμε δείκτες θετικού ισοζυγίου, εάν δεν υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που θα ακολουθούν τα κριτήρια και θα τα κάνουν σεβαστά. Αντιπαραγωγικό επίσης μου φαίνεται να στοχεύσουμε αποκλειστικά και μόνο στις πρασινότερες των πρασινών επιχειρήσεις. Γιατί έτσι αποκλείουμε δυναμικό επενδύσεων ενώ θα έπρεπε να δώσουμε κίνητρα για κάθε είδους επένδυση θα έκαναν οι επιχειρήσεις. Μεθοδολογία. Οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Αλλά και οι κανόνες που θα πλασιώσουν τη μεθοδολογία αυτή πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι, ώστε να μην παρεμποδίζουν την κοινοτομία. Κλείνοντας, επιμένω πως πρέπει να δείξουμε και φιλοδοξία αλλά και ρεαλισμό. Η μετάβαση προς πιο αηφόρο οικονομία είναι μακρύς δρόμος και γι' αυτό χρειάζεται τόσο φιλοδοξία όσο και ρεαλισμός. Ευχαριστώ πολύ, Σάντερ Λούνς, ECR. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα ε, ζητεί συγγνώμη και η Winsborn που δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, εκπροσωπώ εγώ λοιπόν ε, με τις παρατηρήσεις της προς την εισηγητήτρια. Ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή του προβλήματος του greenwashing, τα κοινωνικά ζητήματα και ε, τη διάκριση τους από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πολλά θετικά βλέπει στην έκθεση κυρία Winsborn λοιπόν. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία δεν έχει πιστεί ακόμη από κάποιες τροπολογίες και το λέει αυτό διότι θεωρεί ότι θα μπορούσαν και να επηρεάσουν ακόμη και αρνητικά το συνολικό στόχο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ακριβών και ευρέως χρησιμοποιούμενων οροσίμων. Πρώτον, λοιπόν, θέλουμε η συγγύτρια να διευκρινίσει τις θέσεις της, ε, όπως τις έχει εκφράσει το άρθρο στο ινατροπολογια 13, ε, την ε, απέτηση να έχουν θετικό ισοζύγιο ανεξαρτήτως χρονικού πλαισίου για όλους τους δείκτες την κρίνει πολύ αμφίβολη και επίσης πολλές αμφιβολίες έχει για την τροπολογία 18. Ανταγωνισμός δηλαδή στον τομέα των ε, οροσίμων με την εισαγωγή τελών που έχει συστηθεί επίσης επί μακρόν στις πρόσφατες συνομιλίες για τον κύριο κανονισμό για τα ορόσημα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναρχίσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Επιπλέον επιφυλάξει έχει ως προς τον προσδορισμό της ορολογίας για την αναθεώρηση και την χρήση του όρου πραγματικό κόστος, πράγμα το οποίο ε, θεωρεί ότι δεν εκφράζει σωστά την ιδέα του τέλους, εάν στηρίζεται μόνο σε πραγματικό κόστος. Τρίτον, όπως είπε και η του ΕΛΚ, το ECR θα ήθελε ε, μια πιο ευέλικτη προσέγγιση ε, για το ορόσημα Έχουμε κάνει άλλωστε και όλη τη συζήτηση για τη Συμφωνία για το Κλίμα των Παρισίων. Είναι πολύ σημαντική, ναι. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουμε ότι και η Επιτροπή έχει ε, ανησυχίες και φοβάται ότι εάν συνδεθούν τόσο στενά τα δύο ζητήματα θα είναι πολύ δίσκαμπτο το σύστημα. Άλλο επίσης εκπομπές, άλλο εξοικονομήσεις. Η ΚΕ είναι πολύ επιφυλακτική σε αυτό. Μια προσέγγιση ε, μονολυθική θα περιορίσει και την ε, ποικιλία των πηγών και τη δυνατότητα μέτρησης του ε, αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, οι τροπολογίες 9 και 14 έχουν μια θετική προσέγγιση. Η εισηγήτρια μας λέει ότι θα πρέπει να στηρίζονται στο βαθμό με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός ορισμένων εκπομπών και ότι αυτό θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε όλη την νομοθεσία. Οπωσδήποτε και περιμένει τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους λοιπούς σκιώδης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους λένε. Ευχαριστώ αγαπητή Τζιλ, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης. Χαίρομαι που ε, στηριζόμαστε τους ίδιους στόχους για βιώσιμη, ε, βιώσιμη χρηματοδότηση και βιώσιμη μετάβαση. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όμως ο κόσμο ε, των δικτών αναφορά είναι πολύ περίπλοκος, όπω και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. χωρί του δείκτε αναφοράς, πολλές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα ήταν σήμερα πολύ πιο δαπανηρέ και θα Ω Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά τη νομοθετική ρυθμίση αυτών των δικτών αναφορά. Ήδη στον κανονισμό για του δείκτε αναφορά έγινε πολύ προεργασία. αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα είδο ε, σφραγίδα έγκριση ένα σήματο, ώστε να δώσει σε αυτού που έχουν θετικά κριτήρια αντίκτυπο άνθρακα ούριο άνεμο και μία όθηση. Και συμφωνώ με, τη, με τον προσανατολισμό τη συγγήτρια. Βέβαια, θα πρέπει να κάνουμε κάποιε διευκρινήσει. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον προαιρετικό χαρακτήρα τη ε, νομοθεσία. Επίσης, ε, είναι ζωτική σημασία να αφήσουμε κάποια περιθώριο για διαφορετικές μεθοδολογίες. Το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να φημώσουμε ή να παρεμποδίσουμε την καινοτομία. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό στους στόχους μας για βιώσιμη ανάπτυξη και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες θα βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, διαφάνειας και της συνοχής αλλά και της ελαστικότητας που ε, στηρίζει την καινοτομία. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε για τους πράσινους, η κυρία Μόλι Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ. Η πρόταση φυσικά είναι τμήμα πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μιλήσουμε για τη δημοσίευση, για την νομοθεσία περί δημοσιεύσεων πληροφοριών. Πάντως, το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτεται στο περιβαλλοντικό τμήμα, στο θέμα της βιωσιμότητας και στους σχετικούς δείκτες. Θέλουμε να προωθήσουμε τις φορολοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι καλό βήμα πριν περάσουμε σε δείκτες ε, καλύτερης βιωσιμότητας. Ε, βέβαια υπάρχουν κάποιες ε, συγχύσεις, κάποιο μπέρδεμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τις ε, ε, δημοσιεύσει. Προτιμώ την έκθεση τη κυρία Γκίλ. Χαίρομαι πάντως που ήδη έχει ξεκινήσει την προεργασία η κυρία Νίνα Γκίλ και προσβλέπω στις ε, συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών να ενισχύσουμε περαιτέρω την πρόταση εν ώψη και του τριμερούς διαλόγου. Ε, σίγουρα η ιδέα αυτών των θετικών κριτηρίων για το αντίκτυπο άνθρακα είναι κάπως οξύμορη, γιατί σαν να υπονοούμε ότι υπάρχει κάτι θετικό σε σχέση με το αντίκτυπο άνθρακα, να θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θα έλεγα να το προ... αναφέρουμε ως δείκτης αναφοράς βιωσιμότητας και αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα πράσινο θύλακα, να οθήσουμε όλε τι εταιρείε να ευθυγραμμιστούν το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου του Συμφωνία των Παρισίων και να ε, προβαίνουν σε αιτήσει μειώσει των εκπομπών άνθρακα. Θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία και περιμένω να το συζητήσουμε και με του άλλου σκιώδει ηγητέ. Χαίρομαι που η η Swinburne ε, είναι η σκιώδη ε, των μεταρρυθμιστών συντηρητικών για το θέμα αυτό, γιατί θα μα επιτρέψει να είμαστε ε, συνεπείς και με τον γενικό κανονισμό για τους δείκτες. Δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά παρεμβατική Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε να ρυθμίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια για τις εταιρείε για να μπουν στο, ε, στους δείκτες. Καλύτερα να έχουμε μία προσέγγιση με βάση άδειε για να ε, αποφασίζουν οι επιχειρήσεις τι δείκτε θα υιοθετούν και η Επιτροπή αν πληρούν οι δείκτε τα κριτήρια. Αντί δηλαδή να επιβάλλει τη μεθοδολογία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύτερα να εγκρίνει τι μεθοδολογίε, αφήνοντα ε, ελεύθερο περιθώριο στον ιδιωτικό κλάδο, κάτι που βρίσκεται ακόμη πιο πέρα από την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογή των κατεξιοδότηση πράξεων, ιδιαίτερα στο θέμα τη μεθοδολογία και προτείνουμε σαφή και στενή ευθυγράμμιση με το σύνολο του κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κανέναν από την ΚΟΕ, ούτε από το ΙΕΝΕΦ. Η κυρία είναι στη γενική συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας κλέψω ένα λεπτό, γιατί τα θέματα των δικτών αυτών και της βιωσιμότητας είναι λένεται Στην έκθεση πρωτοβουλίας υπήρχε διακομματική προσέγγιση υπέρ της διεύρυνσης της ιδέας των δικτών, ε, ώστε παράλληλα με τα οικονομικά λογιστικά να έχουμε και κάποιους δείκτες που υπολογίζουν τη βιωσιμότητα της διαχείρισης των πόρων, την κατανάλωση των υλικών, το ύδατος, εκπομπές ε, υπό το πρίσμα της βιοπικιλότητας και ούτω καθεξής καθώς ε, και το Τμήμα Περιβάλλον Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Αν ε, σκεφτούμαστε μόνο με γνώμονα το περιβάλλον, θα καταλήξουμε σε κάποια παράδοξα όπως είχαμε πρόβλημα στη Φιλανδία. Ίσως ε, αποβούμε εις βάρος της βιοπικιλότητας, όπως έγινε με την περίπτωση του Φινικέλεου. Δεν θα πρέπει να ε, επικεντρωνόμαστε μόνο στο περιβάλλον. Και δεν θέλω αυτή να είναι η μοναδική μας ε, έμφαση. Και ελπίζω και ο εισηγητή για τι δημοσιεύσει να αυτή την ίδια προσέγγιση. Θέλουμε ευθυγράμμιση των διαφόρων κανονισμών για να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του και να το λάβουμε υπόψη στους δείκτες αναφοράς. Οι δείκτες θα πρέπει πάντα τα ορόσημα να περιλαμβάνουν τους βασικούς δείκτες για να είναι βιώσιμοι και να μην περιορίζονται μόνο στο κλίμα. Και θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία πώς θα τους υπολογίζουμε τους διάφορους δείκτες. Εγώ θα ήμουν υπέρ της ευελιξίας. Το θέμα είναι να εφαρμόζουμε την αρχή της μη βλάβης, no harm principle. Δεν θα πρέπει ε, ε, το περιβάλλον να είναι εις βάρος ή να παραβλάπτει την ασφάλεια, τη βιοασφάλεια, τη βιοπικιλότητα ή άλλους τομείς. Τι εννοώ λοιπόν. Δεν θέλουμε ξεχωριστό χαμηλό δίκτυ για μικρή χρυσή άνθρακα. Το θέμα των πλούτων, ε, του, της διαχείρισης των πόρων να υπάρχει σε όλους τους δίκτες και να μην περιοριστούμε μόνο στην περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την Τζίνα για το σχέδιο έκθεση. Ένα σύντομο σχόλιο, γιατί και εγώ είμαι συγγήτρια ε, για το επίπεδο 2 benchmark και γι' αυτό με ενδιαφέρει και αυτή η πρόταση. Από το 2020 ε, οι δείκτες αναφοράς ε, θα ρυθμίζονται και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μένα, για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη χαιρετίζω την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει το ε, πλαίσιο σε ό,τι αφορά του ε, δείκτε αναφορά χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσα. Στις επόμενες εβδομάδες θα εργαστώ από κοινού με του συναδέλφου για να διατηρήσουμε το χαρακτήρα του κανονισμού με σκοπό τη διαφάνεια και με γνώμονα την αγορά. Θα καταθέσω όμω και κάποιε τροπολογίε που ήδη έχω καταθέσει στην προηγούμενη αναθεώρηση. Το βασικό σημείο για μένα είναι ότι οι κρίσιμοι δείκτες αναφοράς, όπως το Euribor και άλλοι, έχουν, όπως ξέρετε, σε αυτούς δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε την με του 2020. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να μπορούν να μας εξηγήσουν λίγο παραπάνω το σημείο αυτό. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι μια μεγαλύτερη ε, μεταβατική περίοδος δύο ετών είναι το κατάλληλο μέτρο για να υπάρχουν λιγότερες ε, ταραχές ε, στην αγορά. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Τώρα. Ε, yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Για αυτό το τελευταίο σημείο κατανοούμε ότι υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος για τους κρίσιμε σημασία δείκτες αναφορά των επιτοκίων που μπορούν να παρατεθούν κατά δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι ένα-δύο τέτοιοι δείκτε αναφορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρί περαιτέρω διαδότηση και καθώ η Επιτροπή και η ΕΚΤΕ είναι σε κοινή ομάδα εργασία για εναλλακτικά ε, ενεργοτικού συντελεστέ overnight, εξετάζουμε το ενδεχόμενο παράταση, ούτω ώστε αυτοί οι νέοι ε, δείκτε, εναλλακτικοί δείκτε να μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την αγορά και από τη CCP. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε όλα αυτά για τα παράγωγα, για αυτούς τους νέους δελεστές. Ε, κάτι τώρα επί της σύγχυσης για τις δύο κατηγορίες δικτών, δείκτε αναφορά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και δείκτε αναφορά θετικού αντικτύπου άνθρακα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο παραπάνω ενδεχομένω οι δείκτε αναφορά θετικού αντικτύπου είναι λίγο πιο πράσινοι από του άλλου. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι και οι άλλοι βέβαια. Απλώ ε, με του δείκτε αναφορά θετικού αντικτύπου σημαίνει ότι αφαιρούμε περισσότερο ε, άνθρακα από ό,τι εισάγουν οι άλλοι τρόποι παραγωγής. Όχι απλά περιορίζεται λοιπόν ε, το οικολογικό αποτύπωμα, αλλά αφαιρεί ε, περισσότερο διεξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, από ό,τι ε, εισάγεται από τους ε, εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής. Και έχουμε λοιπόν τους πλέον πράσινους δείκτες αφορά με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Η εισηγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλια. Ευπρόσδεκτα όλα. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί στενή συνεργασία στις συνεδριάσεις των σκιωδών την επόμενη εβδομάδα για να διευθετήσουμε όλα τα ζητήματα που είναι κρεμή και που έχετε επισημάνει. Για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, δεν θα ε, διέλθω όλα τα ζητήματα που ετέθησαν. Όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζουν, την τρίτη η Σύντομα όμως και συνοπτικά. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας έχει ένα πολύ, πολύ καλό ιστορικό και επιδόσει, έχει κάνει αλλαγές στο παρελθόν, στο status quo, σε πολλούς τομείς και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε θετικά και να προχωρήσουμε. Ξέρω ότι πάντα όποτε είχαμε εισαγάγει νομοθεσία ακολούθησε και ο κλάδος ο παραγωγικός, επομένως νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλώς, ευχαριστώ, 24 Οκτωβρίου τροπολογίες, 19-20 Νοεμβρίου εξετά στην Επιτροπή, το Δεκέμβριο στην Ολομέλη. Ευχαριστώ και πάω στο επόμενο, λίγο πολύ το ίδιο θέμα. Πολτάν με κίνδυνο βιωσιμότητα στις επενδύσεις. Τέσσερα 4 λεπτά. 5 πρόεδρε. Καλά. Ε, κάποια λεφτά έχω εντάξει. Και ευχαριστώ βεβαίως ε, το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα στηρίζεται στην έκθεση πρωτοβουλίας που υιοθετήθηκε στο, από το Κοινοβούλιο το Μάιο εφέτος με τη Μόλι Σκοτ και στόχο την ενσωμάτωση των αηφόρων των βιώσιμων επενδύσεων υπάρχει ήδη μία πράσινη προσέγγιση, αλλά θέλουμε αυτό να γίνεται παντού και πάντα. Θέλουμε να ανοίξουμε λοιπόν το πεδίο και πέραν των κεφαλαιοχικών αγορών, κεφαλαιακών αγορών, να το επεκτείνουμε και στις τράπεζες και, και όχι μόνο για πελάτες, αλλά για τον κάθε έναν, όχι μόνο για το κέρδος δηλαδή, αλλά για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη. Αυτά ως γενική προσέγγιση. Πάνω στην έκθεση πρωτοβουλίας χτιζόμαστε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι προθέσεις για την προώθηση αυτή σε παιδοκοινοβουλίου. Ε, πολύ χρήσιμη και επικοδομητική πιστεύω θα είναι και στις συνεδρίες των συντονιστών. Για την ίδια την έκθεση 245 οι τροπολογίες. Καλή η 85, Μακάρτι και Πιέτη Κάινεν για τη συμπερίληψη όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αφού ο στόχος του Κοινοβουλίου είναι να έχουμε το δυνατόν ευρύτερο πεδίο κάλυψης να μην αποκλείσουμε τίποτα και κανένα να είναι ισότιμο το πεδίο για όλους και με ευελιξία. Πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και το να κερδίσουμε την υποστήριξη των τραπεζών. Έχουμε τροπολογίες 55, 53 καρτί, 85 της μόλι, 52 για τον συντονισμό με τη δουλειά που γίνεται στην ε, CRDCRR και θα επισημάνω ότι όταν κάνουμε την αξιολόγηση του κινδύνου, ε, την εισάγουμε νομοθετικά η, ε, ο κλάδος στο, στο, επενδύσεων μας ζητεί διευκρίνεια. Χρειάζεται λοιπόν ασφαλεία δικαίου και αυτό είναι απαραίτητο. Και βλέπουμε ότι και οι πράσινοι με την 111, η με την 112, το ΕΛΚ με την 150 βλέπουμε να υποστηρίζουν τον ίδιο στόχο. ή 128 ή 130 τρεμόσα διευκρινίζουν ζητήματα δέουσας επιμέλειας στη δε αμοιβή. Η βασική αρχή είναι αυτό που λέμε να το κάνουμε, έστω και να μας κοστίσει. Έχουμε λοιπόν ένα 50% της αμοιβή σε μη χρηματοοικονομικούς στόχους, όπως ορίζει και ο σχετικός νόμος των κατοχωρών. Αυτό σημαίνει πληρώνω με βάση αυτά τα οποία έχω υποσχεθεί. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με λύσεις της ε, νομοθεσίας κατηγορίας ε, τομέα 1 και όχι 2. Αυτά ευχαριστώ πολύ για την ε, συνεργασία την επόμενη εβδομάδα και με μια πίεση χρόνου γιατί δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε. Προχωρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάινεν, Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ με σχόλια και ευχαριστίες και προς τον ε, Πρόεδρο της Επιτροπής και προς τους συντονιστές. Έχουμε λοιπόν τη δική μας έκθεση τροπολογίες, αλλά έχουμε και τις άλλες εκθέσεις που, είναι, που αφορούν την, ε, την, ενημέρωση και, την, ε, και τα ορόσημα. καλό θα ήταν λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μια κοινή βάση. Να υπάρχει αυτή η συναντήληψη σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας και να μην προ, χωρούμε με διαφορετικές, ε, ε, με διαφορετικές βάσεις και άρα και διαφορετικές κατευθύνσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και αυτό ήθελα να επισημάνω. Δεύτερον, συμφωνώ ότι πρέπει τη δουλειά μας να τη στηρίξουμε στην έκθεση πρωτοβουλίας και βιβλίο, βέβαιως αυτό ισχύει για, και για τις τρεις εκθέσεις. Αφού υπάρχει ευρύτατη συνένεση ότι οι δείκτες στόχο έχουν να μετρούν τις συνέπειες το εις των επιχειρήσεων είτε είναι οι επενδυτές είτε είναι οι ε, τράπεζες τις οποίες αφορούν οι επενδύσεις. Αυτή είναι η νέα κατεύθυνση. Δέουσε επιμέλεια. Ίσως χρειαστεί μια δουλίτσα εκεί. Δέουσε επιμέλεια και για τις διαδικασίες πρέπει να κοιτάξουμε αλλά και ε, έτσι ώστε να δέσουμε το, κίνη, το κείμενο κατά τρόπον ώστε να μην εκθέσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ε, να μην τις υποχρεώσουμε δηλαδή να αποκαλύπτουν στοιχεία αδυναμίας δικά τους. Σημεία ευάλωτα αυτά πρέπει να παραμένουν ε, απόρριτα για την ίδια την εταιρεία. θέματα που αφορούν δηλαδή, το περιβάλλον και κοινωνικά θέματα. Επίσης, πιστοτικά ιδρύματα και για λόγους ασφάλειας πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, πιστεύω, για το πώς προσφέρονται οι πληροφορίες, οι γνωστοποίησεις, αλλά ταυτόχρονα στα όρια θα πρέπει να κοιτάξουμε να διευκρινίσουμε με βάση τον ε, κανονισμό για την κάλυψη. Αμοιβή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το επίπεδο φιλοδοξίας του συναδέλφου. ώστε να συνδυάσουμε την πολιτική αμοιβών με την βιωσιμότητα. Είναι υπερβολικό αυτό, για να το δε... θα είναι δύσκολο να το δεχθούμε. Για μας αυτό, ως προειδοποίηση ότι εκεί εντοπίζουμε τις κύριες δυσκολίες. Παραρτήματα επίσης έχουμε και έτσι ναι με τους δείκτες είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζουμε τους κινδύνους εκεί που υπάρχουν πράγματι αλλά θα πάμε να διευκρινίσουμε κάθε σημείο μέτρησης πώς δεν είμαι βέβαιη ότι πρέπει να δουλέψουμε με αυτό το επίπεδο εξειδίκευση. Μάλλον χρειάζεται να μείνουμε σε πιο γενικό επίπεδο. Επίσης, ε, ίσονα ζητήματα των ορισμών και άλλα που δεν αφορούν τους επενδυτές. Γιατί δεν θέλουμε να ανατρέψουμε τις ισορροπίες ή να ε, ταλαιπωρήσουμε με υπερβολική λεπτομέρεια στις ε, γνωστοποιήσεις και τη λογοδοσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Χωσάντερ. Ε, θα μιλήσει για το ECR ε, η Λίβ Βίργινη για τους φιλελεύθερους. Αγαπητέ Πολ, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, γνωρίζουμε τις θέσεις σημαίνει τον ΔΕ και έχουμε προχωρήσει διαπραγματεύσεις. Βέβαια, μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ μας. Πιστεύω όμως ότι έχουμε κοινούς στόχους. Βιώσιμη μετάβαση προς βιώσιμη χρηματοδότηση που θα τροφοδοτεί μια βιώσιμη οικονομία. Σε ό,τι αφορά την επέκταση του πεδίου σε όλα τα προϊόντα, με προβληματίζει η προστιθέμενη αξία που θα έχει σε σχέση με το μεγάλο κόστος. Δεν είμαι πεπισμένη ότι το πεδίο εφαρμογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βάλει τα βιώσιμα προϊόντα σε δυσμενή θέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και των επενδυτικών φορέων. Συμφωνώ μαζί σας για τις επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά τα εταιρικά δάνεια δεν νομίζω ότι έχουν, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στον πυρήνα της πρότασης, δηλαδή να αποτρέψουμε την ψευδοοικολογική ταυτότητα. Ούτε πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε συζητήσεις που έχουν γίνει σε θέματα πολιτικής αμοιβών στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Στόχος του κανονισμού είναι να διευκρινίσει κάποια πράγματα, όχι να δημιουργήσει ε, ή να παρεμποδίσει την ασφάλεια δικαίου. υπερβολική φιλοδοξία θα παρεμποδίσει τη μετάβαση που είναι απαραίτητη. Είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε ένα μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους η μόλις, Σκοτ Κάτω. Ευχαριστώ. Καταρχήν είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένη με την εξέλιξη των θέσεων μα για τα βιώσιμα οικονομικά και κυρίω για τα θέματα των γνωστοποιήσεων ή δημοσιεύσεων, αποκαλύψεων. Με σόκαρε στην αρχή όταν ξεκίνησε τη συζήτηση πόσο ελάχιστα γνωρίζουν οι πολίτε ε, πώ κάνουν τι επενδύσει στα επενδυτικά και στα εξοδοτικά ταμεία. Γιατί θα πρέπει να το ξέρουν, είναι δικαίωμά του στου πελάτε. Και όταν υπάρχει τέτοια γνώση και πληροφορία, νομίζω ότι θα ε, τους επιτρέψει να, να επενδύσουν ε, σε εταιρείε που κάνουν πραγματικά βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε για τις διάφορες θέσεις και να προχωρήσουμε στη συζήτηση και στις προτάσεις πριν το διάλογο. Παρόλο που δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία, συγχαρητήρια, Πολ, για τη φιλοδοξία σου να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, ε, ξεπέρασες ε, το πράσινο και το καθαρό ε, τμήμα και ζητάς ε, ε, διαφάνεια για όλα τα προϊόντα και όχι μόνο για τα προϊόντα του στενού τμήματος του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι υπέρ τη βιωσιμότητα και του θεματολογίου για τα βιώσιμα οικονομικά και τη βιώσιμη χρηματοδότηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται, συμπεριλαμβάνονται με την πρόταση του κανονισμού με την πρόταση του εισηγητή, μάλλον και οι τράπεζε. Συμφωνούμε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφεί ποια προϊόντα θα καλύπτονται και να είμαστε ρεαλιστέ ό,τι αφορά το κατόφλι και την περίοδο σταδιακή εισαγωγή. Σημειώνουμε πρόοδο στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κανένα δύο σημεία που χρήζουν περαιτέρω ανάλυση εν ώψη τη ε, συνεδρία τη επόμενη εβδομάδα. Οι πράσινοι πιστεύουν ότι ε, θα πρέπει να έχουμε σαφή ενημέρωση για του συστηματικού κινδύνου μη βιώσιμων επενδύσεων και η πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπο των επενδυτικών του επιλογών. Αυτό όμως, ε, είναι δύο διαφορετικοί στόχοι. Προ το παρόν φαίνεται ότι είναι ε, μπερδεμένοι μεταξύ τους, κάτι που ίσω υπονομεύσει τη θέση του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο. Επίσης, ε, προτάσεις ε, κεφαλαϊκών ε, απαιτήσεων περιλαμβάνουν κάποιες υποχρεώσεις ε, ενημέρωσης. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις διάφορες προτάσεις ενισχύοντας τη φιλοδοξία μας. Θέλουμε μια φιλόδοξη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να περάσουμε στον τριμερή διάλογο ελπίζοντας να μην προδώσει τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και το λαό της Ευρώπης το Συμβούλιο με τις θέσεις του. Ευχαριστώ. Άρκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσει από μένα. Η πρώτη αφορά τη διεύθυνση περιφαρμογή τη πρόταση ε, για να καλύψουμε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεύτερον, έχουμε πρόσθετου ε, κανόνε ε, για σκοπού δέσου επιμέλεια. Κατανοώ ότι θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, ιδίω σε αυτό το θέμα και να καλύψουμε τις, τα αιτήματα για περισσότερε πληροφορίε από τον κλάδο, όμω πρέπει να μετρήσουμε και τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Επιπέρα στο διοικητικό άκθο για μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και αυτό θα αυξήσει και το οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις χωρίς να συμβάλλει ε, σε, στη βιωσιμότητα. Επιπλέον, μια σειρά κράτη-μέλη και η Μάλτη χώρα μου βασίζονται ε, στις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις για υπηρεσίες που δεν αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Πρέπει λοιπόν η εισαγωγή νέων κανόνων για την τόσο επιμέλεια να ακολουθείται και από μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στον εισηγητή. Πολ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ευρεία στήριξη και για την ε, έκθεση πρωτοβουλίας στην οποία βασιστήκαμε. Το βλέπω και από το ΕΛΚ και από τους ε, πρασίνους. Παρότι υπάρχει διχογνωμία, το οποίο εντάξει με δυσκολεύει λίγο, αλλά είπε και η Λίβε ότι θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή και να ε, ακολουθήσει τη θετική ερμηνεία και αυτή νομίζω θα είναι και η βάση είναι και η βάση των συζητήσεων σκιωδών μέχρι τώρα και θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων και στο μέλλον. Προφανώς και με τη δέσο επιμέλεια δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ε, το εμπορικό απόρριτο των επιχειρήσεων, είναι σαφές. συμφωνούμε ότι η μορφή της χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να επιβάλλει και τις απαιτήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι αφετηρία για την ε, εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Ίσως το ίδιο ισχύει και για τον, ε, τον ορισμό των ε, κινδύνων. Αυτή τη στιγμή δεν ορίζουμε τον κίνδυνο, απλώς λέμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι κίνδυνοι, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δεν λέμε όμως ε, πώς θα πρέπει να μετράει κανείς τον κίνδυνο και κατανοούμε ότι πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά, ακόμα και μετά την υιοθέτηση αυτής της νομοθετικής πράξης. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε. Για να απαντήσω έτσι στη ΣΥΡΠΑ, αλλά και στη ΛΥΒΕ, για τον δανεισμό εναντί των επενδύσεων. υπάρχει και μία ακόμα αρχή στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Το είπε και η Λίβε. Θέλουμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο να καλύπτει και να διασκεδάζει αυτέ τι ανησυχίε. Αυτό ισχύει και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σωστά η Μόλι είπε ότι χρειαζόμαστε πληροφορίε, σωστή ενημέρωση και των καταναλωτών, των πελατών. Για να εκφράζουν και εκείνοι τι προτιμήσει τους και όταν έχουν επίγνωση να μπορούν να κάνουν και την αλλαγή. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Σάντ. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι κάτι το καινούριο. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, στα Γαλλία και στις κατοχώρες υπάρχουν ε, νέες προσεγγίσεις εχμής που ήδη υλοποιούνται από ασφαλιστές, από τράπεζες κτλ. Γι' αυτό λέμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά την Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν είναι λοιπόν κάτι το καινούριο. Βέβαια κατανοούμε ότι χρειάζεται χρόνος για αυτή τη μετάβαση. είναι σημαντική μετάβαση, γιατί έχεις δίκιο. Πρέπει... Είναι τράπεζε πολύ σημαντικέ για την χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Ωραία, δεν έχω χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα, επόμενη συνεδρία συντονιστών. Ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφορία προβλέπεται για τις 5 ε, Νοεμβρίου. Θα ήθελα να πω και στη ΣΥΡΠΑ ότι πράγματι θα ήταν χρήσιμο οι συντονιστές να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης ε, και εξέταση των θεμάτων ε, συνέπειας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν. Φυσικά η κάθε ομάδα ε, ενεργεί αυτονόμως και μετά θα τα δούμε εδώ. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία που χρήζουν βελτίωση. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ. Δεν ξέρω κάποιος αντιπρόεδρος θα μπορούσε να συμβάλλει, να σας βοηθήσει και έτσι να διευκολύνει το έργο σας για τις επόμενες εβδομάδες. Ας περάσουμε τώρα στην, στο σχέδιο έκθεσης ε, της ΕΚΤ για το 2017 του κ. Γκαμπριέλ Μάτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την πρώτη συνάντηση των σχεδόν ηγετών για να εκπονήσουμε συμβαστικές τροπολογίες. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Λάθος σειρά. Διάβασα. Το θέμα της πολιτικής ανταγωνισμού το αναβάλουμε για άλλη φορά. Ήταν να εισηγητήσω με ο κύριος Ρεμόν ή ο Σβέν Κίγκολτ. Συγγνώμη, ξεπεράσαμε, ε, το προσπεράσαμε. Λυπάμαι, λυπάμαι. Ε, Νομίζω ότι θα έχεις αποφασίσει να το αναβάλουμε, αλλά δεν ε, το έκανες. Θα διαβάσω λοιπόν εκ μέρους του εισηγητού, Μισελ Ρεμό, που δυστυχώς στέλνει τη... ζητά συγγνώμη γιατί κολλείεται σήμερα. Φυσικά περιμένει στενή συνεργασία με τους και συγγετές προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπημένη συμβαστική πρόταση και είναι, θα είναι στη διάθεσή τους πολύ γρήγορα προκειμένου να συζητηθούν οι προτεραιότητές σας και περιμένει και φυσικά και τις τροπολογίες σας. Όπως ξέρετε λοιπόν, η πράσινη είναι γενικώ υπέρ ε, καλών επιδόσεων στον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα η κοινή αγορά ε, χρειάζεται αυστηρούς ελέγχους και στα θέματα του ανταγωνισμού και του θεμητού ανταγωνισμού, ισότιμου ανταγωνισμού. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε το ε, ακαθόδε ζήτημα των ε, φορολογικών επιδοτήσεων και των επιλεκτικών πλέον εκτιμάτων στον τομέα αυτό. Θεωρούμε ότι η φετινή έκθεση για τον ανταγωνισμό στάθηκε κυρίως σε τρεις προτεραιότητες ε, και εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατρανώσουμε τη φωνή μας ε, χωρίς να καλύπτουμε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, αλλά να επικεντρωθούμε σε τομείς όπου ο πολίτης πιστεύει πως η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να τύχει κάποιες επανισορρόπησης. Οπότε, η πρώτη πρόκληση είναι η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας. Και η ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών φέρνει νέες ευκαιρίες ε, και προκλήσεις με τα δεδομένα να είναι ο βασικός φορέας της οικονομικής ισχύω. Οι επιχειρήσεις χαρά, σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με στόχο και με χαμηλή τιμή να συγκεντρώσουν όσο περισσότερα δεδομένα γίνεται από τους χρήστες. Και ε, ουσιαστικά από τη στιγμή που έχουν τον de facto έλεγχο των δεδομένων αποκλείουν τους αντιπάλους τους ε, από την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Κάτι που δημιουργεί εμπόδια για τους καταναλωτές και προβλήματα πρόσβασης ε, στα καινοτόμα προϊόντα της επιχειρήσης και της υπηρεσίας. Οι εταιρείε αυτές πολύ συχνά επιβάλλουν ε, άδικες ε, συμβατικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, με τη μορφή ευρέων αδειών για την συγκέντρωση δεδομένων σε χρήστες που μάλλον δεν θα αλλάξουν παρόχους. Κάτι που δημιουργεί μεγάλους φραγμούς και εμπόδια. Ε, σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση τη πολιτική ανταγωνισμού την εποχή τη παγκοσμιοποίηση ψηφιοποίηση, η έκθεση υποβάλλει σημαντικέ εκθέσει και προτάσει. Θεωρούμε ότι ο έλεγχο δεδομένων είναι ένα δείκτη τη ε, αγορά ισχύω με βάση το άρθρο 102 τη Συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πρόσφατη μεταρρυθμίση του αντίστοιχου γερμανικού νόμου και μάλιστα σημαντικές υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας θα πρέπει να απαιτούνται μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και των παρόχων ε, δικτύων, ε, κοινωνικών δικτύων. Και για να αποφύγουμε περιπτώσεις όπως ε, συγχώνευση του WhatsApp και του Facebook, θα πρέπει να εξετάσουμε πιο στενά τα κατόφλια που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση του ελέγχου της συγχώνευσης στις ε, αξίες της, ε, στην τιμή της ε, οικονομίας της αγοράς που εκπροσωπείται μερικές φορές από τον αριθμό των επισκεπτών σε συγκεκριμένη στο σελίδα. Επίσης, και τα εμπόδια για την εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία είναι πολλές φορές ανυπέρβλητα, στο μέτρο που αυτή η άδικη συμπεριφορά διονύζεται. Τόσο πιο δύσκολο είναι να καταπολεμήσουμε τέτοιες αντι, ανταγωνιστικές συμπεριφορές και αποτελέσματα κατά του ανταγωνισμού. Το είδαμε με την υπόθεση της Google. Τη μέχρι ότου ληφθεί η απόφαση, οι περισσότεροι ανταγωνιστές είχαν ήδη εξωθηθεί, ε, ε, παραμεριστεί από την αγορά. Ε, ο εισηγητής θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά ενδιάμεσα μέτρα, με προσωρινά μάλλον μέτρα, και να προσπίσει τις, ε, τα δικαιώματα ταυτόχρονα των εταιριών που βρίσκονται υπό έρευνα. Θέλουμε ε, τη θεωρία της ε, μη βλάβης και δεν επικεντρώνεται μόνο στην τιμή, αλλά και σε μη χρηματοοικονομικά θέματα, όπως είναι η ιδιωτικότητα των πολιτών. Το δεύτερο μείζον θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε είναι ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν ε, μπορεί να λαμβάνει δράση χωρίς να λαμβάνει υπόψη και άλλους τομείς της ευημερία των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την αλυσίδα ανεφοδιασμού σε τρόφιμα, μας ε, θορυβεί η μεγάλη συγκέντρωση που υπάρχει στον τομέα αυτό, με ολέθρια αποτελέσματα για τους γεωργούς, τους καταναλωτές, το περιβάλλον, αλλά και την καινοτομία σε τελική ανάλυση λόγω του περιορισμού του ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε την ε, συγχώνευση Μονσάντο και Μπάγερ παρόλο που είπε ότι η απόφαση της ε, προσδιορίζεται και κατοχυρώνεται από τις, συνθήκε συνθήκες και την ε, πιστιστική ασφάλεια ή την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ο κανονισμός περί συγχωνεύσεων με τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί ε, στόχους δημοσίου συμφέροντος στη διαδικασία ελέγχου των συγχωνεύσεων. Κάτι που αυτή τη στιγμή μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Χίγκολτ. Ναι, τελειώνω. Και ενώ το δίκαιο ανταγωνισμού και η εφαρμογή του δεν περιορίζουν την υπερβολική ε, εξουσία στην αγορά, τα πολλά καρτέλ ε, με βάση το άρθρο 101 έχουν ε, αντιμετωπιστεί ως εμπόδιο στη συνεργασία μικρών φορέων της αγοράς ε, που τηρούν περιβαλλοντικά και Πρέπει να κλείσετε όμως τώρα, φτάνει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτεραιότητες για την έκθεση και την επανεξέταση της ε, ε, νομοθεσίας για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ, Χόκμαρκ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ μέσω του κύριου Γκίγκολτ, τον εισηγητή. Για την πολύ καλή δουλειά και εγώ προσβλέπω σε καλές ε, συζητήσεις, παρατηρήσεις τώρα. Βεβαίως όλοι ζητούν ανταγωνισμό μέχρι ότου τον βρουν. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναστήσουμε μια συνολική προοπτική γιατί η δυναμική της, πολι... της, οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηριχθεί στον ανταγωνισμό, εξαρτάται από τον ανταγωνισμό. Από εμά εξαρτάται λοιπόν να τον ε, διευκολύνουμε με τρόπο επακριβή αλλά και χωρίς περιστολές Πρέπει να ανοίξει η αγορά και βέβαια έχουμε να κάνουμε εδώ με μια προσέγγιση κέρια σημασία που θα ορίσει και το πώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Μπορούμε ή να ρυθμίζουμε τις υφιστάμενες οντότητες ή να αφήσουμε ανοιχτό πεδίο για την είσοδο νέων παραγόντων. Και να αφήσουμε να ορίσει ο ανταγωνισμός τη σημασία που θα προσλάβει ο καθένας. Εδώ λοιπόν βλέπω πόσο λάθος ή πόσο σωστά μπορεί να κρυθούν αυτά τα πράγματα. Νομίζω και τις δύο λύσεις πρέπει να ε, δεχθούμε, τα παράλληλα να τις προωθήσουμε, γιατί ούτε η μία ούτε η άλλη μπορούν να αποκλειστούν. Ε, μία αξιολόγηση σε σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες είναι απαραίτητα ή... Είναι απαραίτητο λοιπόν το και σημαντικό να τονίσουμε ότι πολλές είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν ανοίξει, είτε πρόκειται για ταξίδια, είτε για πολλά άλλα τεράστιο τομέα υπηρεσιών. Είναι πολύ η παράγοντες που έχουν ε, δραστηριοποιηθεί και τα επίπεδα βέβαια, ο όγκος των συναλλαγών που δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει πριν από 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι υπάρχει διευκόλυνση στον ανταγωνισμού σε πεδίο πολύ ευρύτερο από ό,τι θα μπορούσαμε πριν από 10 χρόνια να υπολογίσουμε. Δεύτερον, το πιο σημαντικό είναι να αφήσουμε ένα πεδίο για την ανάδειξη νέων πλατφορμών οι κοινωνικές πλατφόρμες για τις οποίες συζητούμε σήμερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες που συζητούμε σήμερα, μπορεί να έχουν μόνο ιστορία 10 ετών, προσφέρουν όμως μεγάλο η υπηρεσία στον καταναλωτή Ο κατακαιρματισμός λοιπόν προκειμένου να στηριχθεί ένας ε, ανταγωνισμός ε, δεν είναι απαραίτητο ότι εξυπηρετεί τον ε, καταναλωτή. Και μπορώ να πω ότι σε 10 χρόνια θα μιλούμε για άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όχι αυτές που συζητούμε σήμερα. Καθήκον μας λοιπόν είναι να αφήσουμε πεδίο ανοιχτό για νέες οντότητες που θέλουν να αναδειχθούν. Φορολογία και τραπεζικά. Πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι φορολογικοί, οι πολιτικοί και οι κανόνε που θα σαχθούν να μην επηρεάσουν τον ανταγωνισμό, δηλαδή να μην σχεδιαστούν έτσι ώστε να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Σε αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και επακριβεί. Τράπεζε. Έχουμε περιθώριο για κρατικές παρεμβάσεις με τους κανόνες που έχουμε και νομίζω ότι μπορεί το κοινοβούλιο να το διαφυλάξει αυτό. Πρέπει να τελειώνεται όμως. Ναι, εκεί που δεν βλέπω όμως αναφορά είναι τα θέματα της ενέργειας. Καλώς ευχαριστώ και όλα αυτά τα της Gazprom. Αλλά υποτάσσομαι στις ε, επιθυμίες σας ε, κύριε Πρόεδρε και σταματάω εδώ. Κύριο Σάνιε. Πρόεδρε ευχαριστώ. Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιώδους σημασία εργαλείο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα την Επιτροπή με την Επίτροπο Βέστακερ η οποία έχει εξασφαλίσει τόσα θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ανταγωνισμού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω μία από τις θετικές πρωτοβουλίες των σοσιαλιστών δημοκρατών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα αποτελεσματικότητας για το μέλλον, δηλαδή την επιβολή στις αρχές, εθνικές αρχές ανταγωνισμού, μια διαδικασία που έχει φτάσει πια στον τριμερή διάλογο μετά την έκθεση πρωτοβουλία που είχα εγώ συντάξει το 2016 και όπου έλεγε ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν πρέπει να ανατρέπουν κοινωνικά επιτεύγματα μπορούμε να κάνουμε πολλά σημαντικά και με την αυτή πρόταση πιστεύω και φέτος. Ο κύριος Χαϊμάν νομίζω έχει κάνει αυτό που όφιλε με την έκθεσή του. Μπόρεσε να εντοπίσει δηλαδή με όλους τους περιορισμούς στην έκταση της έκθεσης τα ζητήματα τα σχετικά με τον ανταγωνισμό που έπρεπε να ε, φυγούν και επιβεβαιώνω χωρίς να επισέρχομαι σε λεπτομέρειες ότι και η ομάδα μου πιστεύει πως πρέπει να στηρίξουμε θέματα περιβάλλοντος και ανταγωνισμού ιδιαίτερα και να εξασφαλίσουμε ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας. Βεβαίως αντίρρηση δεν έχουμε για τη συμπερίληψη και θεμάτων ενέργειας που ανέφερε ο κύριος Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθούν οι προτεραιότητες μας όπως τις αναφέρει η έκθεση για την καινοτομία, τις ποιοτικέ θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη της επενδύσης, την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση της ενίας αγοράς και ιδιαίτερα την ψηφιακή και ενεργειακή ενιαία αγορά. Πριν από δύο χρόνια το είχα αναφέρει, το επαναλαμβάνω, ότι χρειάζονται περισσότερα βήματα για την ενίσχυση τη ε, εσωτερική αγορά, τη ενιαία αγορά μέσω μια φορολογική ένωση, η οποία θα εξασφαλίσει ισότιμου όρου στην ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα, Πρόεδρε, θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει του κανόνε και τι διαδικασίε που θα ισχύουν για τι κρατικέ ενισχύσει στον τραπεζικό τομέα και πριν ε, προχωρήσουμε στην διατύπωση των περαιτέρω τροπολογιών ή μέχρι τη διατύπωση των περαιτέρω τροπολογιών. Θέλω να επισημάνω πως το Κοινοβούλιο πιστεύω πρέπει να έχει εξουσίες και συναπόφασης στην πολιτική αυτή, στην πολιτική του ανταγωνισμού. Για άλλη μια φορά λοιπόν ζητούμε την αναθεώρηση προς την κατεύθυνση αυτή των συνθήκων Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδους ε, εισηγητές για ένα καλό κείμενο το οποίο θα συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις. Στόχος μας οπωσδήποτε πρέπει να είναι μόνο η διευκόλυνση της καθημερινής ζωής του πολίτη αλλά και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ Σανταλούς από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος δεν μπορούσε να δώσει σήμερα. Ο Ρόμπερτ Σιλίπε. Ε, χαιρετίζει τι προσπάθειε του εισηγητή για την έκθεση. Δύο παρατηρήσεις έχει μόνο. Ο Σκιώδη από πλευρά CCR ε, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονό ότι ο εισηγητή ε, επικεντρώνεται περισσότερο σε κλαδικέ ανεπάρκειες και δεν κατανομάζει συγκεκριμένε επιχειρήσει. Ο Ρόμπερ θεωρεί και συμφωνώ ότι έτσι είναι ε, πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη η έκθεση. Επικεντρώνεται στα συστημικά προβλήματα. Είναι θετική η πρόταση ε, για τις ε, αιτήσει εκθέσεις. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι και μια ε, σειρά άλλοι κλάδοι παρουσιάζουν τέτοιες πρακτικές, τέτοια φαινόμενα και θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών, για γέννη και στα συνδρομικά δίκτυα, όσο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, και στο πλαίσιο του κλάδου της ενέργειας, όπου ανέφερε και ο συνάδελφο, μιλήσατε για τον αθέμητο ανταγωνισμό, τι πρακτικέ ε, στον τομέα του φυσικού αερίου και από προσωπική άποψης είναι σημαντικό να μην γίνει μια έκθεση επί της φορολογίας, αλλά επί του ανταγωνισμού. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο. Ε, πολύ θετική λοιπόν η προσέγγιση του έγινε αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια ξεκάθαρη συζήτηση και μετά για την παράγραφο 9 Ήταν και μια τροπολογία που είχα καταθέσει εγώ πέρυσι. Είχα μια συζήτηση με την κυρία Βερστάγκερα αν πρέπει να εξετάσει ε, τον ε, ε, επιβαρυντικό παράγοντα και αντίκτυπο της ποσοτικής χαλάρωσης. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και σήμερα. Εκτιμούμε λοιπόν το γεγονός ότι και σε ψηλότερο επίπεδο πλέον θα γίνει αυτή η συζήτηση. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν προς τον εισηγητή των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω άλλους κοιόδης. Ε, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Κάρλες Μόσο, για ορισμένε παρατηρήσει, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δυστυχώ θα πρέπει να σα ζητήσω να, είστε, ε, να συντομεύετε, γιατί έχουμε και άλλο σημείο στη μέση Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς τον εισηγητή αρχικά για το σχέδιο έκθεση και προς ε, την Επιτροπή στο σύνολό τη ε, για την στήριξη ε, που επιδεικνύεται για, την, για ένα εύρωστο σύνολο κανόνων. Πολύ σωστά, η συγητή επικεντρώθηκε σε μια σειρά βασικών προτεραιοτήτων. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που παρουσιάζει η ψηφιοποίηση στην πολιτική ανταγωνισμού. Βέβαια, έχουμε και ευκαιρίες μαζί με τους κινδύνους. Ήδη λαμβάνουμε υπόψη στην, στον τομέα της εφαρμογής ζητημάτων που πάνε πέραν ε, των ανταγωνιστικών τιμών, για παράδειγμα πώς οι συγχωνεύσεις μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση των δεδομένων το πρόσφατο παράδειγμα της Apple και του Shazam ε, με δευτεροβάθμια ε, συνέχιση της έρευνας είναι ένα καλό παράδειγμα σε τη φορά την χρήση δεδομένων στις πλατφόρμες. Θέλουμε να είμαστε ε, στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτηση, Γι' αυτό και η Επίτροπος κυρία Βερστάγκερ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μία και θα συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της τον του χρόνου και θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση. Έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση με πάνω από 100 ε, συμμετοχές από τον κλάδο και είναι πολύ θετικό που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να αλλάξουμε το, το σύνολο κανόνων ή τον τρόπο που εφαρμόζονται. Το δεύτερο που αναφέρατε είναι ο αντίκτυπος ορισμένων πρακτικών στο περιβάλλον. Σε ένα βαθμό, σίγουρα και στην, στον τομέα της επιβολής του νόμου όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη Μίλησατε για την εξέταση της περίπτωσης Bayer Monsanto, μία από τις περιπτώσεις πέρσι στον αγροχημικό κλάδο, όπου επικεντρωθήκαμε όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στον αντίκτυπο ε, στην καινοτομία. Που, καινοτομία που θα μας ε, έδινε καλύτερα ή ασφαλέστερα προϊόντα για το περιβάλλον. Και εμείς επιβάλλουμε ε, σημαντικά έχει αγγεία σε αυτή την επιχείρηση, ώστε να μην περιοριστεί η καινοτομία σε αυτόν τον κλάδο. Και έτσι να έχουμε καλύτερα προϊόντα στο μέλλον. Όπω ανέφερε και η Επίτροπο στην παρουσίασή τη, πρέπει να διακρίνουμε του τομεί όπου η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί όντω ε, να κάνει τη διαφορά από του τομεί όπου το κανονιστικό πλαίσιο μα δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Ε, η ύπαρξη με την ύπαρξη δικτών αναφορά, καλύτερο είναι να ε, ακολουθήσουμε την άκουσα του, του κανονιστικού πλαισίου. Μένω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ σύντομα, κύριε Γκέκολτ. Καταρχήν ευχαριστώ το ΕΛ και το ECR που επισήμαναν το θέμα της ενέργειας. Και εμείς έχουμε πρόβλημα με κάποια συμπεριφορά που είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό και μας, προ... μας ανησυχεί. Και χαίρομαι που το συζητάτε και ελπίζω να μας στηρίξετε σε... στα θέματα της τρέβλους ανταγωνισμού λόγω εξωτερικών παραγόντων των εκπομπών διοξιδίου του άθρακα που πραγματικά στρεβλώνουν ιδιαιτέρως τον θεμητό ανταγωνισμό στην ενεργειακή αγορά γιατί ε, τα εξωτερικά αποτελέσματα το, της πυρηνικής ενέργειας ή των ορυκτών καυσίμων δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές τουλάχιστον σε αποτελεσματικό επίπεδο. Άκουσα με ενδιαφέρον ε, αυτά που είπατε, Γκούναρ, για τις πλατφόρμες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πολύ συχνά οι πλατφόρμες ε, ανοίγουν αγορές εκεί που δεν υπάρχουν ουσιαστικές αγορές. Δεν είμαστε κατά των πλατφόρμων, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε πολλές ε, αγορές έχουμε ε, μονοπόλια και ολιγοπόλια, κάτι που οδηγεί είτε σε κλείσιμο των αγορών ή σε χειραγώγηση των αγορών. Και μπορεί να γίνει και κατάχρηση α, της α, δεσπόζησης ισχύω. Και εμεί είμαστε υπέρ των μικρών ξενοδοχείων και είμαστε κατά τις επιβαρύνσεις, κατά 15% του τζίρου τους από το booking.com και άλλες πλατφόρμες που κάνουν τις κρατήσεις γιατί αυτή η προστιθέμενη αξία ανήκει στις περιφέρειες. Τέτοιου είδου χρεώσεις λοιπόν, τέτοια τέλη δεν θα πρέπει να συνιστούν το κογλυφία. Γιατί μερικές φορές είναι τόσο υψηλά που ισοδυναμούν με το κογλυφία. Επίσης, θα πρέπει να αναλύσετε τις συνέπειες που θα έχει η συγχώνευση της Μπάγκερ με τη Μοσάντο σε άλλου τομεί. Έχουμε και άλλο σημείο, λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε άλλο σημείο. Δυστυχώ η ερμηνεία προβλέπεται μέχρι τις 12.30. Ε, Η 26 Οκτωβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες, 19 Νοεμβρίου συζητάμε και ψηφίζουμε αργότερα. Περνάμε στην έκθεση του Γκαμπριέλ Μάτο, πολύ σύντομα, και περνάω στα, αγγλικά, ε, στα ισπανικά. Ε, είχαμε την πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πολύ επικοδομητικά δέχτηκα 230 τροπολογίες. Δεν είναι πολλές, αλλά μερικές φορές ε, είναι αντίθετες. Ήθελα να κρατήσω θετική γραμμή σε ό,τι αφορά το έργο της ΕΚΤ και την παρούσα κατάσταση. Ε, είναι πολύ σημαντική ενέργεια τα τελευταία χρόνια και οι οικονομίες της αγοράς σε ένα μεγάλο βαθμό χάρη στην ε, πολιτική του Νομισματικό Ταμείο και τη διαρθρωτική πολιτική που έχουν ε, προωθήσει ορισμένα κράτη-μέλη. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και δείχνουν ε, μια ανάπτυξη πέραν του 2% και ποσοστό ανεργίας 7%. Επαναλαμβάνω πολύ θετικό, όπως ε, επαναλαμβάνω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Brexit, λαϊκισμός, προστατευτισμός είναι η κίνδυνη σε σχέση με την δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν οι στόχοι της αποκατάστασης της, ε, των επενδύσεων που είναι ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ σημαντικές. Και βεβαίως συμφωνούμε απολύτως για όλες τις πτυχές μιας πολιτικής επεκτατικής